Θα θέλουμε να καλωσορίσουμε την Ελένα Εσπινόζα, Υπουργό Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Θαλασσίου και Φυσικού Περιβάλλοντος και την καλωσορίζουμε για να μας κάνει μια εισήγηση. Αγαπητή Ελένα, αυτή είναι η πρώτη προεδρία που αρχίζει υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας, που εισήγαγε σοβαρές αλλαγές ε, για την ΚΑΠ. Με την συναπόφαση, με την ε, τακτική διαδικασία της ε, συναπόφασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα φέρουν εξίσου την ευθύνη στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας και γι' αυτό θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις που σχετίζονται με την παρούσα συγκυρία. Γι' αυτό, αγαπητή Ελένα, προτείνω στο μέλλον να έχουμε πάντα έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου στις ε, συνεδριάσεις μας της Επιτροπής Γεωργίας και υπαίθρου έτσι ώστε να είμαστε κοινωνοί των αλλαγών και των εξελίξεων στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Εμείς αναμένουμε πολλά από την Ισπανική Προεδρία, από τη δική σας Προεδρία και από το ρόλο του Συμβουλίου. Και σήμερα θα αντιμετωπίσουμε μαζί το θέμα της ΚΑΠ μετά το 2013 μέχρι το 2020 και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και του τομέα γεωργίας και τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το ρόλο των γυναικών στις αγροτικές περιφέρειες. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόντες και δίνω το λόγο στην Ελένα Εσπινόζα που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας. Σε ευχαριστώ Ελένα και έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι ενώπιόν σας για να σας μιλήσω για το πρόγραμμα εργασίας για την ΚΑΠ κατά την Ισπανική Προεδρία. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, γνωρίσαμε πολλές θεσμικές αλλαγές, ιδιαίτερα σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην συναπόφαση. Θα ισχύσει λοιπόν η διαδικασία συναπόφασης και για την ΚΑΠ. Όπως, όπως ανέφερε και ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Θαπατέρο, θα συνεργαστούμε στενά και σίγουρα οι αποφάσεις θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα και θα βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Θα σας ορίσω τις προτεραιότητές μας στον τομέα της γεωργίας εντάχει έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμμεριστούμε απόψεις και να υποβάλλετε και ερωτήσεις. Για μας η γεωργία και η πολιτική τροφίμων είναι στρατηγική τομής για την Ευρώπη. Για να μπορέσουμε να προμηθεύουμε τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς με ε, τρόφιμα σε καλές τιμές και ποιοτικά προϊόντα και αυτό στα πλαίσια του νέου οικονομικού μοντέλου βιώσιμης οικονομίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να συνεισφέρουμε στην ε, τήρηση των στόχων της χιλιετίας. Θα έχουμε τρεις προτεραιότητες. Το μέλλον της ε, ΚΑΠ πέρα από το 2013, την υποστήριξη της ε, γεωργικής και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανίας τροφίμων και την ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στο αγροτικό περιβάλλον. Το μέλλον της ΚΑΠ πέρα από το 2013 αποτελεί προτεραιότητα για την Ισπανική Προεδρία έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αυξήσει την παραγωγή προς μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αγορά. Γι' αυτό χρειάζεται και μια κοινή αγροτική πολιτική που να είναι ιδιαίτερα ε, δυνατή και ευρωστή. Δεν ε, πρέπει να αποδομήσουμε τις κοινέ πολιτικές που αντικατοπτρίζουν τους στόχους της συνθήκης κατά ικανοποιητικό τρόπο. Ούτε η Προεδρία μπορεί να ε, αποτολμήσει κάτι τέτοιο. Η ΚΑΠ αποτελεί έναν πύχη σταθερότητας, μια σταθερά. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχει την κατάλληλη δημοσιονομική πρικοδότηση. Έτσι θα μπορέσει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Το θέμα του μέλλοντος του, της ΚΑΠ δεν είναι καινούριο. Είχε αρχίσει πριν από το, τον υγειονομικό έλεγχο, όπως όρισαν και οι προγενέστερες προεδρίες. Η Ισπανική Προεδρία θα προσπαθήσει να εξεύρει τα κατάλληλα μέσα διαχείρισης της αγοράς και διαχείρισης κρίσης, που είναι μέσα απαραίτητα για την βιωσιμότητα της ΚΑΠ. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανίας τροφίμων. Θα προωθήσουμε τις επενδύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή, διευρύνοντας τις αγορές μας. Θα πρέπει να προωθήσουμε τα προϊόντα μας σε τρίτες χώρες, και να υπάρχει αμοιβαιότητα απαιτήσεων σε σχέση με ασφάλεια και ποιότητα καθώς και την ε, ευημερία των ζώων. Ένας άλλος στόχος της Προεδρίας είναι η βελτίωση της λειτουργίας της διατροφικής αλυσίδας, έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με βάση όλους τους κρίκους της διατροφικής αλυσίδας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής θα προσπαθήσει να βελτιώσει τη διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη. Ο τομέας τροφίμων αποτελεί το 2% του κοινοτικού ΑΕΠ και αποτελεί το 13,5% της συνολικής απασχολησιμότητας του μεταποιητικού, τομέα. Έχουμε 300.000 θέσεις εργασίας και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις κρίσης καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Τη στιγμή που θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη διεθνή κρίση, πιστεύω ότι θα είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί, θα δημιουργούμε απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε και τα σύνορά μας έτσι ώστε να προμηθεύουμε και τρίτες χώρες. Το τρίτο κατά προτεραιότητα στοιχείο είναι ο ρόλος της γυναίκας στον αγροτικό κόσμο. Ο αγροτικός κόσμος, ο αγροτικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από γύρανση, από παρουσία ανδρών, από υψηλές τεχνολογίες και από τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Η Προεδρία θεωρεί αναγκαίο να προωθήσουμε ευρωπαϊκές πολιτικές ισότητας έτσι ώστε να επιβιώσει ο αγροτικός ιστός, κάτι το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς τις γυναίκες. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε άλλα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού που θα έχουν και σοβαρές επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα. Πρόκειται για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την ε, απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τους υποκείμενους όρους, με τους όρους που διέπουν αυτή την πολιτική. Επίσης θα προστατεύσουμε τα ζώα και θα προωθήσουμε θέματα ευζοίας. Θα δώσουμε συνέχεια στις εργασίες δηλαδή που είχε αναλάβει η Σουηδική Προεδρία με την οποία εργαζόμαστε. Όπως θα δείτε, ένα εξάμεινο γεμάτο προκλήσεις που ελπίζω ότι θα διεξαχθεί σε ένα πνεύμα συνεργασίας και θετικού συντονισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που έχουν σε μάσα ο τομέας των γεωργών και οι πολίτες της Ευρώπης, γυναίκες και άνδρες. Σας προσφέρω τη δική μου συνεργασία εγώ προσωπικά. Την συνεργασία μου ως <clears throat> Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προεδρεύουσα και όλης της ομάδας μου μια κοινή τέτοια εργασία και συνεργασία θα κάνει μια πιο δυνατή Ευρώπη, πιο κοντινή στους πολίτες, αλλά επίσης και με ένα τομέα όπως τον τομέα της γεωργίας που θα τον τονώσουμε και θα πετύχουμε πολλούς στόχους ελπίζω όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Έλενα Σπινόζα, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σου μια ισχυρή ΚΑΠ για το μέλλον. Όχι η διάλυση. Είναι θέματα τα οποία ήδη έχουμε αντιμετωπίσει στην ακρόαση με τον νέο επίτροπο που κάναμε πριν λίγες μέρες. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Θα έλεγα ότι ε, κάνει ομοιοκαταληξία με τη λέξη αμοιβαιότητα. Εμείς είμαστε υπέρ τη ασφάλεια τη διατροφικής, προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα μάλιστα ασχοληθήκαμε με τη γεωργία και τις κλιματικές αλλαγές, αλλά χρειάζεται αυτοί οι κανόνες να γίνουν σεβαστοί και από τις χώρες που εξάγουν. Είναι πολύ σημαντικό και είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ανταγωνιστικότητα αυτό. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν για την εισήγησή σας και ξεκινάμε τη συζήτηση ε, με, τον, με την κυρία Ελίζα Ελιζαμπέτα. Α, η Άννα είναι η πρώτη. Μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Υπουργό διότι μας εξέθεσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας διότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις αλλά ελοχεύουν και πολλοί κίνδυνοι. Όπως είπε και ο πρόεδρος ε, ο κ. Ντεκάστρο συναντηθήκαμε με τον ε, υποψήφιο επίτροπο και μας είπε ποια είναι, ποιο είναι το νέο όραμα της γεωργικής πολιτικής όπως ελέγχθηκε από την κυρία, προελέχθηκε από την κυρία Φίσερ Μπόουλ. Υπάρχουν ε, δύο ζητήματα, ή συμφωνίες με τρίτες χώρες και ιδιαίτερα η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου, η οποία συνήφθη ορισμένες εβδομάδες πριν. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες, υπάρχει μεγάλη ε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη που διέπει αυτό το σύστημα διότι δεν υπάρχει σωστό καθεστώς αμοιβαιότητας με τις ε, τρίτες χώρες. Και οι ποσοστώσεις που ε, ορίζονται πλήττουν χώρες της Νοτιού Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ισπανίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ποια θα είναι η, η θέση μας διότι εμείς ταχθήκαμε κατά αυτής της συμφωνίας, διότι αντιβαίνει και ε, πλήττει την κοινοτική παραγωγή. Θα πρέπει δηλαδή να εξεύρουμε μέσα έτσι ώστε τρίτες χώρες να τηρούν τις ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες. Θα πρέπει να υπάρχουν συστηματικοί έλεγχοι, διότι πολλές φορές τρίτες χώρες δεν ε, τηρούν τους όρους των συμφωνιών. Ένα άλλο θέμα είναι το μέλλον της ε, ΚΑΠ. Από το Υπουργείο μας ε, δώσατε ένα έγγραφο και χαιρόμαστε διότι υπάρχει μια θέση, σε, υπάρχει θέση για ορισμένα θέματα, αλλά η συγχρηματοδότηση δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι υποχρεωτική μετά το 2013. Πολλοί θέλουν επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, διότι η γαλλική κυβέρνηση ανέφερε το γεγονό ότι η κυβέρνηση Σαρκοζή αντιτίθεται σε οποιαδήποτε συγχρηματοδότηση μετά το 2013. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα μίας ευρωπαϊκής δασονομικής πολιτικής, διότι σήμερα το πρωί μιλήσαμε για θέματα περιβάλλοντος και δεν μπορούμε να παραμείνουμε με την ανακοίνωση κατά της ξηρασίας, διότι δεν προβαίνει στη σύσταση μιας πραγματικής δασονομικής πολιτικής, δασικής πολιτικής. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι αγροτικές οργανώσεις και ενώσεις ε, μιλούν υπέρ ενός εισοδήματος, εγκυμένου εισοδήματος. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με ένα ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, όπως το ορίζουν και ε, ασφαλιστικές εταιρείες. Τι θα γίνει με το εγκυμένο εισόδημα στην ΚΑΠ. Ο κύριος Σαντός, Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντά σας και εξ ονόματό μου και εξ ονόματο τη ομάδα μου θα ήθελα να εκφράσω τις ε, επιθυμίες για την πιο επιτυχή ολοκλήρωση της Προεδρίας σα. και έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτήν εμεί Φυσικά και επειδή δεν είναι συνηθισμένο. Έχουμε μία υπουργό, υπουργό Γεωργίας ταυτόχρονα και υπουργό περιβάλλοντο. Ξεχωριστό αυτό η απόφαση να σας διορίσει υπουργό και για τη γεωργία και για το περιβάλλον προβλέπει μια πολύ σωστή διασύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και γεωργίας. Φυσικά έμεινα πολύ ικανοποιημένο με τις προτεραιότητες που μόλις μας διαβιβάσατε. Για όλους εκείνους που είναι υπέρ μιας ισχυρής ΚΑΠ στην Ευρώπη να ακούσει κανείς ότι η γεωργία και τα θέματα των τροφίμων είναι στρατηγική σημασία και το περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές όπως και σήμερα το πρωί είχαμε ευκαιρία να συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε σε σχέση με μια έκθεση που συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον συνάδελφό μας Στέφαν Φολ και που καταδείχθηκε με επαρκώς ισχυρό, ε, ε, εντυπωσιακό τρόπο την ανάγκη να ενταχθεί στην μελλοντική ΚΑΠ αυτή η συνιστόσα των κλιματικών αλλαγών με συγκεκριμένους χειροπιαστούς όρους και όχι μόνο θεωρητικά. Και έτσι λοιπόν και για την ίδια την απασχόληση. Η θέση απασχόλησης πρέπει να είναι μια σταθερή συνιστόσα για να νομιμοποιείται σωστά η ΚΑΠ. Σε αυτό ακριβώς θέλω να θέσω ερώτημα. Εμείς έχουμε τεράστια πρόκληση και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται στα επόμενα δύο χρόνια μέχρι ότου ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Τα δύο κέρια θέματα θα είναι ο προπολογισμό, αλλά για τον προπολογισμό δεν θα πω τίποτα, δεν θα τοποθετηθώ. Επειδή είπε και η Υπουργό ότι η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν επαρκή κονδύλια για την ΚΑΠ. Όμω είναι αναγκαίο να καθορίσουμε πρώτον το πρότυπο τη γεωργική πολιτική που επιθυμούμε. Και αυτό σε σχέση με το πρότυπο, το πιο σημαντικό θέμα είναι η βάση του κριτηρίου των άμεσων ενισχύσεων και αυτό μετά το 2013 με την αποσύνδεση από την παραγωγή είναι αδύρυτη ανάγκη να εξεταστεί. Και εδώ λοιπόν σε σχέση με τις απόψεις και ιδέες ε, που εκφράζονται, σε σχέση με ένα κριτήριο για μια πιο δίκαιη και πιο εξισορροπημένη ΚΑΠ μεταξύ των περιφερειών, των γεωργών και των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι το λόγο τώρα έχει ο George Lyon. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω την Υπουργό και τι παρατηρήσει τη, την εισήγησή τη, ιδιαίτερα τη δέσμευσή τη για μια ισχυρή κάπα καθώ και για τα όσα είπε για τη βιωσιμότητα της γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εγώ θέλω να μιλήσω για ένα από τα θέματα κλειδιά που ανέφερε ε, για την Προεδρία, ότι δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στην αγορά, όπου έχουμε πολύ μεγάλη πτητικότητα, ιδιαίτερα στον τομέα του γάλακτος, που μόλις ε, ξεπεράσαμε μια πολύ, πολύ μεγάλη κρίση με χαμηλές τιμές. Πιστεύετε ότι πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα από την κρίση του γάλακτος και τι ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε ώστε να προλάβουμε μια άλλη κρίση. Και η Κομισιόν να ανταποκριθεί με πιο αποτελεσματικό και ταχύτερο τρόπο. από ό,τι την τελευταία φορά. Και Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση του γάλακτος και άλλες κρίσεις που μπορεί να προκύψουν το μέλλον. Ευχαριστώ. Grazie George. Martin Hosling, ναι, κυρία Υπουργέ, και εξ ονόματο τη δική μα κοινοβουλευτική ομάδα σα καλωσορίζω θερμά εδώ ανάμεσά μα. Επιθυμούμε καλή συνεργασία, ε, εξαιρετική συνεργασία μαζί σα και μετά από την πρώτη επαφή μπορώ να πω ότι θέτεται σωστά τα κέντρα βάρους ε, με τον ορθό τρόπο. Αυτό που επιθυμούμε βέβαια είναι, μια και ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή διαδραματίζουμε πλέον έναν άλλο ρόλο, να συνεργαστούμε ενισχυμένα, ενδυναμωμένα. Στην αλυσίδα λήψεων αποφάσεων να εμπλεκόμαστε πλήρω και όχι να μας γνωστοποιούνται κάποιες αποφάσεις εκ των υστέρων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε να υπάρχει μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων στο μέλλον. Είναι πολλά τα σημαντικά στοιχεία που αναφέρατε και σε ένα σημείο σας υποστηρίζω απόλυτα και σας ευχαριστώ που το επισημάνατε τον σημαντικό ρόλο της γεωργίας και του τομέα των τροφίμων για την διασφάλιση θέσεων απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια ίσως αυτό κάπως αγνοήθηκε, αλλά ακριβώς σε περίοδο οικονομικής κρίσης πρέπει να θέσουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το τομέα και όχι να είναι ένας τομέας ο οποίος θα μέσα στο πλαίσιο των ορθολογικών μεταρρυθμίσεων να αγνοηθεί και εξαρτώνται χιλιάδες θέσεις απασχόλησης από αυτόν. Συμφωνούμε μαζί σας. Η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας είναι σημαντικό σπουδαίο εγχείρημα και μέλημα και έτσι η εργασία σε σχέση με την ε, δευτερογενή ακόμα απασχόληση. Ο ρόλος της ε, γυναίκας δεν έχει επαρκώς ακόμα αξιολογηθεί σε αυτά τα πλαίσια. Θα μας ενδιέφερε ως κοινοβουλευτική ομάδα σίγουρα μια και κατά το τελευταίο εξάμεινο ασχοληθήκαμε έντονα με την κρίση για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών, αν έχετε κάποιες νέες απόψεις και προτάσεις να υποβάλλετε, αποκινούμε την ομάδα υψηλών αξιωματούχων, high level group. Η ρύθμιση των αγορών είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εκτός συζήτησης για σας ή υπάρχει δυνατότητα να ξανασυζητηθεί το θέμα για, με ρυθμίσεις για την αγορά. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο δεν αναφέρθηκε ακόμα είναι το ότι βρισκόμαστε στο έτος ε, της βιοπικιλότητας έτσι τους στόχους που θέσαμε εμείς ενώπιόν μας δεν τους υλοποιήσαμε και στη Γεωργία έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Πώς αυτό θα το λάβετε υπόψη στο μελλοντικό σας σχεδιασμό και πώς θα το εντάξετε στο σχεδιασμό σας. Σε ένα άλλο σημείο μπορείτε να πείτε κάτι πιο εξειδικευμένο. Είπατε ότι θέλετε να εξισορροπήσετε τα στοιχεία της αγοράς. Ιδιαίτερα για μας ο ρόλος της Γεωργίας θα πρέπει στην αγορά να ενισχυθεί. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Εμείς ως κοινοβουλευτική η ομάδα έχουμε ήδη μια πρώτη έκθεση σχετικά είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα των επομένων μηνών πώς μπορούμε αυτές τις δυσαναλογίες στην αγορά να τις εξισορροπήσουμε πάλι θα μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις προτάσεις σας τελευταίο θέμα ΠΟΕ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κατά πόσο συμφωνείτε με τις απόψεις του νέου Επιτρόπου ότι εδώ η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επαρκής και δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες υπαναχωρήσεις ευχαριστώ Ευχαριστώ Μάρτιν. Τώρα μετά από αυτό το γύρο εκπροσώπων των ομάδων ξεκινάμε με την Ελίζαμπεθ Γέγκλη. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Προεδρεύουσα, καλώς ήρθατε. Θερμά θέλω να σας πω εδώ στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας σας. Εσείς στο Συμβούλιο παρόμοια θέματα παρουσιάσατε και όλα όσα άκουσα μέχρι στιγμής και διάβασα από τις τοποθετήσεις σας και σε σχέση με την, τον αρμόδιο επίτροπο στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάνουν να σκέφτομαι ότι θα μπορούσατε να έχετε μια καλή ομάδα που θα συνεργάζεται ισχυρά για τα, ε, το άμεσο μέλλον. Αυτή είναι η εντύπωσή μου και παρακαλώ να δώσετε και αυτή τη συνεργασία σε σχέση με εμά. Θα ήθελα κυρίως το θέμα των γυναικών στον χώρο της υπαίθρου να αναφέρω Χάρηκα που αυτό το θέμα είναι μία από τις προτεραιότητές σας ως Ισπανικής Προεδρίας. Όμως πιστεύω ότι με αυτό το σκηνικό δεν πρέπει μόνο τις γυναίκες να λάβουμε υπόψη που εργάζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά τους χώρους της υπαίθρου ως σύνολα. Και να προβληματιστούμε να δούμε πώς για νέες γυναίκες, νεότερες γυναίκες, μπορούμε να δώσουμε ευκαιρίες πέρα από την καθαρή ασχολία και ενασχόληση με τη γεωργία, στον τουρισμό για παράδειγμα, ή σε άλλες δραστηριότητες να τους δώσουμε μία απασχόληση, μία θέση εργασίας συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαι αρμόδια για την ε, Επιτροπή Γεωργίας για την οδηγία δοκιμών όσον αφορά τα ε, ζώα θα ήθελα εδώ να πω ότι έχουμε μια συμφωνία με σχεδόν όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Είχαμε και μια συμφωνία και με τη Σουηδική Προεδρία σχετικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή τη συμφωνία και αυτή τη συνένεση σε αυτό το σημείο πώς την αντιμετωπίζετε εσείς εξειδικευμένα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η εξέτασή του. Ευχαριστώ. Γκαρσία Πέρες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες σε σχέση με την παρουσίασή σας σε αυτή την κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Εδώ και κάποιους μήνες ήδη διεξάγουμε μια συζήτηση εδώ για το ποιο θα πρέπει να είναι το μέλλον και πώς θα το αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την ΚΑΠ. Νομίζω το συμμερίζονται όλοι αυτό το ενδιαφέρον που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α, τώρα πλέον εφ' με τη συνθήκη της Λισαβόνας που αναλαμβάνει θεμελιώδη ρόλο και που θα είναι συμμέτοχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνομοθέτης. Πρέπει να εντείνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συσχετισμό και τις εργασίες και το συντονισμό μεταξύ μας σε σχέση με αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μας κάνατε, παρουσιάζοντας και θέτοντας τη γεωργία ως ένα στρατηγικό τομέα για την ΕΕ. Είναι θεμελιώδους σημασίας τώρα να μπορέσουμε να απαντήσουμε, να δώσουμε απαντήσεις σε εκείνους τους τομείς που διαμφισβητούν την νομιμότητα και την ανάγκη μιας κοινή αγροτικής πολιτικής. Και ένα μέτωπο στρατηγικό που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, τη διασφάλιση των, ε, της διατροφής. Είναι θεμελιώδη θέματα. Και επίσης κάτι άλλο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το έργο που επιτελεί η ε, γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα καθορίζοντας τη δυνατότητα να ζουν στην Ήπεθρο αρκετοί πολίτες. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπουμε ότι αποψηλώνεται πολλές φορές η Ήπεθρος από το ανθρώπινο δυναμικό της, χρειαζόμαστε τη γεωργία για να παραμείνουν οι άνθρωποι σε αυτούς τους χώρους και να αναπτύσσουν εκείνες τις δραστηριότητές τους τους εκείνοι που επιθυμούν να συνεχίσουν να διαβιούν στον χώρο της υπαίθρου. Και τώρα σε σχέση με συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις προτεραιότητες που μας παρουσιάσατε θέλω να σας ρωτήσω πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε την προτεραιότητα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ από το 2014 ως το 2020. Όπως σας είπα είναι συζητήσεις ανοιχτού χαρακτήρα και που διεξάγονται με ανοιχτό χαρακτήρα και όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την δυνατότητα μέσω ακροάσεων να αντιμετωπίσει, να καλύψει αυτό το θέμα. Πώς σκοπεύετε να καλύψετε αυτή την προτεραιότητα πρώτα. Ποιε δραστηριότητε ε, σκοπεύετε να αναπτύξετε για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τη γεωργία και τη ε, ε, τροφικής παραγωγής από πλευράς μας στην Ευρώπη και για τον ρόλο των γυναικών στον χώρο της υπαίθρου. Είναι σημαντικός αυτός ο ρόλος, θεμελιώδης και μέτρα σαν αυτά τα οποία δρομολογήθηκαν από την κυβέρνηση της Ισπανίας σε σχέση με την κοινή συμμετοχή όσον αφορά ε, ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις καταδεικνύουν την πρόοδο για αυτό το σημείο. Η γυναίκα εργαζόταν πάντα στον χώρο της υπαίθρου και στη γεωργία αλλά με αόρατο τρόπο άφαν, άφαντος συμμέτοχος που δεν ήταν διάκριτος ο, ο ρόλος και ο χαρακτήρας του. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν περαιτέρω δράσεις ώστε να τονωθεί αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα έχει το λόγο ο Αντιπρόεδρος Νικουλέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Υπουργέ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και εύχομαι καλή τύχη. Όπως και οι συνάδελφοι που ήδη και εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Υπουργό να μας παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία χειροπιαστά για τον ρόλο της γυναίκας στον χώρο της Υπέθρου. Επειδή 40% των πολιτών μας ζουν στον χώρο της Υπέθρου. και είναι αυτονόητο και ότι έχουμε εδώ ότι πάνω από το ίμιση είναι γυναίκες και έχουμε, αναφέρθηκε η Υπουργό στην υπεργύρανση όσον αφορά τον χώρο τη υπαίθρου. Ερωτώ, έχει η Ισπανική Προεδρία τον στόχο να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα δίνοντα ε, αρρωγή υποστήριξη στου νέου γεωργού. Ευχαριστώ, Μαρτίνε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι οι προτεραιότητες που επεσήμανες αξίζουν την υποστήριξή μας και μεταξύ άλλων είναι συνεκτικές και συνάδουν με τις πολιτικές που αναπτύσσει η χώρα μας που με την κυβέρνησή της συμπίπτουμε πλήρως και αισθανόμαστε ότι μας εκπροσωπεί επαρκώς. Κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν πιο πριν για το θέμα του προϋπολογισμού και των προοπτικών για τη γεωργία, των κονδυλίων και των προοπτικών. Πιστεύω ότι απόλυτα συμφωνούμε με την τοποθέτηση ή αυτά τα οποία απορρέουν ως συμπεράσματα από την παρουσίασή, τους, παρουσίασή σου, ότι δεν είναι αποδεκτό από εμά να μειωθούν τα κονδύλια από πλευράς προϋπολογισμού που θα αφιερώνονται στην κοινή αγροτική πολιτική. Τούτου λεχθέντος πρέπει να δούμε πώς θα το διασυνδέσουμε, πώς θα το παντρέψουμε αυτό και θα το συντεριάξουμε με τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει εμείς οι ίδιοι να κοινοτικοποιηθούν άλλες πολιτικές. Βρίσκεται μέσα στον στόχο μας να μην επαρκεστούμε ότι ουσιαστικά η μόνη πολιτική θα είναι η πολιτική για τη γεωργία που θα είναι κοινοτικοποιημένη ενώ οι άλλες θα είναι εθνικοποιημένες. Θέλουμε να προχωρήσουμε με την κοινοτικοποίηση, όμως να το δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό χωρίς να περικοπούν κονδύλια για τη γεωργία. Αυτό θα μας ε, οδηγούσε ή στη συγχρηματοδότηση, ούτε και με αυτή συμφωνούμε πρέπει να πω, ή στην αύξηση του όγκου του προϋπολογισμού των κονδυλίων που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη οδός για να ολοκληρωθεί η Ευρώπη όπως και αγραφείται και αναπτύσσεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, τούτου λεχθέντος και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά υπάρχουν σημαντικοί τομείς, ισχυροί τομείς ακόμα και χώρες ολόκληρες που θεωρούν ότι το ποσοστό των κονδυλίων που αυτή τη στιγμή αφιερώνονται στην κοινοτική αγροτική πολιτική ε, είναι ε, ε, Δεν συμφωνούμε με αυτό, αλλά μην αγνοούμε ούτε το βάρος ούτε την επιρροή αυτών, κυρίως στην Ευρωβουλή που τώρα θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Το δεύτερο σχόλιο από πλευράς μου, Υπουργέ, έχει σχέση με την κυρίαρχη ε, δραστηριότητά μου στη συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική δράση από πλευράς μας. Πρώτον, όσον αφορά αυτά και κάνοντας λόγο για συμφωνίες όπως αυτές που υπεγράφει με, την, με το Μαρόκο, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ποιο είναι, ποιοι είναι οι κανόνες του θεσμικού μας οργάνου. Το, το, το Κοινοβούλιο δεν τροποποιεί συνθήκες. Το Κοινοβούλιο επικυρώνει ή δεν επικυρώνει συμφωνίες και συνθήκες, αλλά δεν τροπολογεί. Ή λοιπόν πρόκειται για άγνοια ή για δημαγωγία όταν κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τροποποίηση ενώ αυτά δεν μπορούν να τροποποιηθούν από πλευρά μας εξόρισμα Κανοντα Κάνοντας λόγο για αυτά τα θέματα, δεν πρέπει να παραμείνουμε στην ε, επιφάνεια των πραγμάτων επιφανειακά. Δεν μπορούμε να επιθυμούμε να εισάγουμε ή να υπάρχει διευκόλυνση συγκεκριμένου ποσοστού προϊόντων που εισάγονται από χώρες του τρίτου κόσμου και από την άλλη πλευρά, όπως είναι λογικό, αντί ε, για παράδειγμα να έχουμε ντομάτες που θα εισάγονται, να έχουμε σκαφίδια και ε, σχεδίες που θα έρχονται με αυτές οι, μετα, με, οι μετανάστες στις χώρες μας. Πρέπει να δούμε πώς θα συντεριάξουμε αυτά τα δύο πράγματα τα δύο προβλήματα και την παράνομη μετανάστευση και την εισαγωγή και βοήθεια ε, προϊόντων από ε, τρίτες χώρες. Πρέπει να δούμε ότι δρούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία ζητούμε ε, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή τις, την Ισπανία για την πλειοψηφία των προϊόντων που παράγονται από εμά και που τώρα θα εισάγονται από το Μαρόκο στην Ευρώπη. Να δούμε πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει αντιμετωπιστεί. Αυτά ήθελα να αναφέρω πρόεδρε και με παρουσίες σαν τη δική σου εδώ ανάμεσά μας κατανοούν οι συνάδελφοι πόσο σωστή είναι η δράση του Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες θα πατέρω πρωθυπουργού της ε, Ισπανίας όπου εξίσου γυναίκες και άνδρες ε, υπουργοί σε ισότιμο επίπεδο ε, δρούν και εργάζονται για να μην μείνουμε πίσω και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ευχαριστώ Μαρτίνες. Και τώρα ο κύριος Ανιού. Τρεις παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Ε, και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε σε αυτό, όταν σταμάτησε να μιλά η Υπουργό. Ε, δηλαδή, οι αμοιβαίε εμπορικέ συμφωνίε ε, στι παγκόσμιο, παγκόσμιο επίπεδο. Θα το αντιμετωπίσετε σε δύο-τρία χρόνια όπου η Ιταλή και η Ισπανή παραγωγή δεν θα μπορούν να παράγουν αυγά σε συστοιχίε κλοβών. Και οι καταναλωτέ θα θέλουν να τρώνε αυγά και πιθανότατα θα εισάγονται από την Ουκρανία και από την Ινδία. Έτσι όπω έχουν τώρα τα πράγματα στις σχέσεις με τον ΠΟΕ, δεν επιτρέπεται να απαγορέψουμε τη συνεισαγωγή οποιοδήποτε υλικού που βασίζεται απλά με βάση μόνο τη μέθοδο παραγωγή. Με χαρά άκουσα ότι θα το αμφισβητήσετε, αλλά θα ήθελα να ξέρω πώ ακριβώ θα το κάνετε. Δεύτερη παρατηρήση αφορά το ρόλο των γυναικών στην Γεωργία. Τώρα, αυτό είτε είναι μια, ένας ευσεβής πόδος είτε θα βάλετε και κάποια χρήματα στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή οι, οι εργοδότες να παίρνουν κάποια ανταμοιβή αν προσλαμβάνουν γυναίκες ή θα τους αναγκάσετε. Τώρα, ε, παραδοσιακά ε, στη Γεωργία, ιδιαίτερα στην ε, εκτροφή ζώων ασχολούνται, κυρίως στα πουλερικά, αλλά ίσως και στα ζώα. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε ότι δεν οδηγούν καθόλου τα τρακτέρ. Στη Βρετανία, ας πούμε, στις μεγάλες, στα μεγάλα αγροκτήματα όπου οργώνουν με τα τρακτέρ ε, θα επιμείνετε ώστε να χρησιμοποιούν και γυναίκες. Τέλος, για τις κλιματικές αλλαγές. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι όποιες αποφάσεις ληφθούν για αυτά τα ζητήματα θα βασιστούν σε επιστημονικά πορίσματα. Ευχαριστώ. Στεφάν Λεφόλ. Bon, δεν είναι εύκολο να παρέμβει κανεί μετά από τον κύριο Χιούς γιατί έχει έναν ε, ωραίο τρόπο να παρουσιάζει τα πράγματα. Ε, εγώ υποστηρίζω απόλυτα τον στόχο, δηλαδή τη θέση των γυναικών στην Γεωργία και στον κόσμο της υπαίθρου αποτελεί νομίζω και ένα γενικό στόχο της Ισπανικής Προεδρίας. Ε, δεν μπορούμε παρά να τον υποστηρίξουμε. Ε, επίσης, συμμερίζομαι τους στόχους που θεσπίζονται μέσω της ε, ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας, γεωργικής βιομηχανίας. Όπως είπαμε εδώ πρόκειται για πάρα πολλές ε, θέσεις μισθωτών. Επίσης μοιράζομαι την ιδέα, συμμερίζομαι την ιδέα πως πρόκειται για μια ε, γεωργική πολιτική που είναι και διατροφική πολιτική. Αλλά να προσθέσω ένα στοιχείο γιατί είστε ταυτόχρονα υπουργό ε, Γεωργίας και Περιβάλλοντος και Στη Σαραγώσα είχαμε συμμετέχει σε ένα συνέδριο σε σχέση με το πρόβλημα του νερού. <coughs> Η πολιτική, ναι, πρέπει να είναι γεωργική, πρέπει να είναι τροφική, αλλά θα πρέπει για το μέλλον να εντάξει και την περιβαλλοντική διάσταση. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη. αυτό. Επίση, σε επίπεδο της Ισπανικής Προεδρίας θα ασχοληθείτε με το θέμα των μεγάλων προσανατολισμών που μπορεί να προτείνει η Κομισιόν για την περίοδο μετά το 2013 και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε μια γεωργική πολιτική κάπως αναδιοργανωμένη σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα, από ό,τι είδα σε κάποια από τα έγγραφα που αφορούσαν ε, τους στόχους ε, του Ισπανικού Γεωργικού, ε, Υπουργείου Γεωργίας υπήρχαν ιδέες ενδιαφέρουσες για την αναδιοργάνωση του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Μήπως μπορείτε αυτά κάπως να τα αναπτύξετε. Εν πάση περιπτώσει, συμμερίζομαι τους στόχους σας και υποστηρίζω απόλυτα την Προεδρία αυτή και τα όσα θα μας προτείνετε στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ, Στεφάν. Εγώ έχω ακόμα 7 που έχουν ζητήσει το λόγο. Αν τα πείτε πιο γρήγορα θα έχουμε και τη δυνατότητα να ακούσουμε την απάντηση της Ελένα. Ο Ζωζέ Μποβέ. Καλημέρα σας, κυρία Υπουργέ. Έχω τρεις ερωτήσεις να θέσω. Πρώτη είναι συγκυριακή και αφορά την κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρετε πως υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των ε, γεωργών, των αγροτών. Χιλιάδες αγρότες είναι στους δρόμους. Υπάρχουν, ε, έχουν κάνει μπλόκα στα σύνορα διότι οι Έλληνες αγρότες ζουν μια πολύ ε, δύσκολη κατάσταση όπως κι άλλοι την έχουν περάσει αυτή την κατάσταση. Έχετε ήδη στο όνομα του Συμβουλίου αποφασίσει να παρέμβετε σε σχέση με την κατάσταση των Ελλήνων αγροτών. Αν ναι, τι προβλέπετε. Δεύτερο, δεύτερη ερώτηση. Η Κομισιόν ήδη επανελειμμένος και τέλη Δεκέμβριο 2008 ήδη παρατηρούσε ότι το μερίδιο τη προσθέμενης αξίας ε, για τα γεωργικά προϊόντα από το 1975 που ήταν 31% δηλαδή το κέρδος των γεωργών τώρα βρισκόμαστε στο 24% είναι ε, στοιχεία που ήδη έχει θεσπίσει η ίδια η Κομισιόν. Δηλαδή οι αγρότες αμείβονται πολύ χειρότερα και η προστιθέμενη αξία πάει είτε στα, στις ε, εταιρείε διανομής είτε στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό το λαμβάνετε υπόψη και πώς απαντάτε. Τρίτη ερώτηση. Όπως είπε ο συνάδελφος Σλίνγκ. Το 2010 είναι το έτος της ε, βιοπικιλότητας. Και μιλήσαμε για τη βιοπικιλότητα εν γέννη. Εγώ μίλησα για την γεωργική βιοπικιλότητα και σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δυστυχώς ιδιαίτερα στην Ισπανία έχουμε πρόβλημα με τη δυνατότητα των ε, βιολογικών εκμεταλλεύσεων να μπορούν να καλλιεργούν ε, καλαμπόκι, αραβόστο χωρίς να μολύνονται από τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πώς σκοπεύετε να επιβάλλετε το σεβασμό του δικαιώματος να καλλιεργεί κανείς με ή άνευ. Γιατί αυτοί που το κάνουν, ε, σε κάποιες χώρες το κάνουν, αλλά αυτοί που δεν το επιθυμούν τελικά ε, μολύνονται. Ελπίζω πως το 2010 θα είναι όντως μια χρονιά που θα σεβαστούμε αυτούς που δεν θέλουν να μολυνθούν ε, τα αγροκτήματά τους. Ευχαριστούμε, Ζωζέ. Παπαστάμκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την έκθεση των προγραμματικών προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας. Ε, ξεκινώ από εκεί που ε, άρχισε ο, και ο κύριος Μποβέ. Ε, πράγματι προσυπογράφω την περιγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα. Οι αγρότες είναι στους δρόμους ε, και έχουν μπλοκάρει όλες τις εθνικές, όλο το εθνικό οδικό δίκτυο αλλά και συνοριακές πύλες, ιδίως προς βορράν με τη Βουλγαρία, με ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και αυτό δείχνει και την απόγνωση της Ευρώπης της υπαίθρου ε, ε, της, ε, και τα διέξοδα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου, χωρί, ανήκω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι χαμένοι είναι και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές με αυτό το μοντέλο κοινή αγροτικής πολιτικής. Και θα το πω ευθέως, έχω την αίσθηση ότι κερδισμένοι είναι μόνο οι πολυεθνικές ε, αγροβιομηχανιες agrobusiness, όπως επίσης και οι πολυεθνικές αλυσίδες τροφίμων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα δύο ερωτήματα που θέλω να σας κάνω πολύ σύντομα. Η... η Ισπανική Προεδρία σκοπεύει να ενεργοποιήσει μηχανισμούς στήριξης άλλων γεωργικών αγορών, άλλων προϊόντων κατά το παράδειγμα της στήριξης του τομέα του γάλακτος που ήταν ορθή αυτή η στήριξη ε, άλλων ευαισθητών προϊόντων που αφορούν και τη χώρα, αφορούν και τον Ευρωπαϊκό Νότο ιδιαίτερα. Παραδείγματος χάρη ενεργοποιώντα το αποθεματικό το οποίο υπάρχει. Ε, θα ήθελα την άποψή σας από αυτό το σημείο. Ε, το δεύτερο σημείο, εάν φιλοδοξείτε, ω Ισπανική Προεδρία να θέσετε τις βάσεις για την, μετά το 2013, τις βάσεις της συζήτησης για την κατεύθυνση της ΚΑΠ μετά το 2013, τώρα, κατά τη διάρκεια αυτού του, ε, εξαμήνου. Και το τρίτο σημείο υπόθηκε, έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις του γύρου ε, της Δόχα, εάν θεωρείται ως τελειωμένη, ως επαρκή τη διαπραγματευτική προσφορά, το όφερ που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προηγούμενες απόπειρες διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του γύρου της Δόχα ή αν θέλετε, τώρα που αναζωπηρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, να διαμορφωθεί μια άλλη εντολή, ένα άλλο mandate, ένα άλλο μαντά ε, προς την Κομισιόν, η οποία θα φέρει και το βάρος των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κανιέτε. Η κυρία με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, αφήγηση των προτεραιοτήτων. Εγώ προέρχομαι από τη Λετωνία που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση έπρεπε να περικόψουμε 500 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό και έπρεπε να πληγεί ιδιαίτερα η γεωργία και οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Οι αγρότες τώρα στη Λετωνία λαμβάνουν έξι φορές λιγότερο άμεσον, ε, άμεσες επιδοτήσεις σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη. Άρα έχω ένα αίτημα προς την ε, Ισπανική Προεδρία. Οι πρώτες σοβαρές ε, συζητήσεις θα γίνουν επί της Προεδρίας σας σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΚΑΠ. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση δίκαιη κατανομή πληρωμών δηλαδή ίση πρόσβαση στους όρους ανταγωνισμού όλων των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή και σε ένα άλλο ζήτημα. Πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία συναπόφασης για αγροτικά θέματα. Δεν έχει παρέλθει πολύς χρόνος από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και η Ισπανική Προεδρία θα πρέπει να είναι καινοτόμος στη δράση και στις αποφάσεις της. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Άνωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να εισακουστούμε και εμείς. Γίνανε πολλές συζητήσεις σε σχέση με τους πυλώνες της αγροτικής πολιτικής πρόσφατα. Ακούγονται πολλές φήμες ότι τα Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να κινηθούν προς τα περιφερειακά χαρτοφυλάκια για χρηματοδότηση και θα ήθελα τη δική σας γνώμη επί του θέματος. Ευχαριστώ. Σικερέσκι. Σικερέσκι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η, γεωργία στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερα πολλές μορφές, ε, έχει μεγάλη ποικιλία, έχουμε μεγάλες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ε, ανάλογα με το που στρέφεται κανείς ε, στο βορρά ή στο νότο, έχουμε ορεινή γεωργία, έχουμε παιδινή γεωργία και έχουμε διαφορές. Πρέπει εδώ τώρα σε σχέση με την δυνατότητα της ενδιάμεσης αναθεώρησης που διανοίγεται μπροστά μας και της επανεξέτασης ε, τι θα γίνει μετά το 2013 σε σχέση με τα όσα θα διαπιστωθούν από την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, ένα θερμό καλωσόρισμα στην Επίστροπο Εσπινόζα. Πώς να μην συμμεριστεί κανείς ε, τις ε, προτεραιότητές σας. Είναι ουσιαστικές για τις δικές σας ενέργειες και για την Ισπανική Προεδρία για αυτό το εξάμεινο. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη σημαντική δήλωση που κάνατε σε σχέση με τον γεωργικό τομέα λέγοντας πως είναι στρατηγικός ρόλος του. Μιλήσατε για τις, ε, την πολυλειτουργικότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να ξαναδώσουμε στον Γιώργο το ρόλο του που δεν είναι ο να κάνει τον κυπουρό, αλλά ε, εκείνο ο ρόλος του είναι να παράγει γεωργικά προϊόντα, διάφορα. Βιοπικιλότητα. Είναι το Ευρωπαϊκό Έτος της Βιοπικιλότητας. Θεωρείτε, κυρία Επίτροπε, πως ε, ήρθε η στιγμή να ξαναδούμε στο πεδίο της βιοπικιλότητας την 479 ε, του 89 που είναι γνωστή ως οδηγία για τα πτηνά που έχει, είναι μια οδηγία που ε, χρονολογείται πια εδώ και 30 χρόνια. Ήταν λίγα τα κράτη-μέλη τότε. Τώρα υπό το φως της διεύρυνσης σε 27 χώρες ε, μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε εκείνες, ε, εκείνα τα παραρτήματα, να τα ενημερώσουμε και να εγγυηθούμε περισσότερα και καλύτερα με μέσα ε, για τη διατήρηση της ε, πανίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ακόμα σημαντική ερώτηση. Στις προτεραιότητές σας υπογραμμίσατε την υπόθεση της εργασίας των γυναικών, δηλαδή την ευχή να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στη Γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μιας πρωτοβουλίας της ε, αποφάσισε την ακύρωση την ε, κατάργηση του τομέα του καπνού στην Ευρώπη. Και θα μιλήσουμε μετά για αυτή την υπόθεση, γιατί θα παρουσιαστεί μια μελέτη όσον αφορά τον αντίκτυπο της εφαρμογής της κοινοτικής πρωτοβουλίας της Κομισιόν για τον τομέα του καπνού. Λοιπόν, από αυτή τη μελέτη στη σελίδα 15 προκύπτει σαφώς το γεγονός ότι αν όντω εφαρμοστεί αυτή η επιλογή λανθασμένη της ε, Κομισιόν για το τομέα του καπνού θα υπήρχαν ε, αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα της απασχόληση. Και όπως το γνωρίζετε, η μεγαλύτερη η πλειοψηφία μάλλον των γυναικών, ε, μάλλον η πλειοψηφία των εργαζομένων στον καπνό είναι γυναίκε. Αντί να μιλάμε λοιπόν και να δημιουργούμε νέες πολιτικές. Γιατί να μην διασυντηρήσουμε ε, πολιτικές που ήδη υπάρχουν και που εγγυώνται ε, την απασχόληση των γυναικών και που εγγυώνται επίση σημαντικά έσοδα σε οικονομικό επίπεδο. Ποια είναι η δική σα τάση ε, σε σχέση με αυτέ τι προτάσει τη Κομισιόν, προτάσει οι οποίε διεψεύθηκαν τέσσερι φορέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σε μεγάλη πλειοψηφία επανέλαβε την βούληση που υπάρχει οριζόντια σε όλε τι πολιτικέ ομάδε να μην εκμηδενήσουν τον τομέα του καπνού, αλλά να εγγυηθούν όπω και σε όλε τι άλλε γεωργικέ παραγωγέ ένα αξιοπρεπέ μέλλον μέχρι το 2013 και πέρα από αυτό. Ποια είναι η δική σας θέση, ε, Υπουργέ. Ευχαριστούμε κύριε Μπερλάτο, δεν μπορούμε παρά να συμφωνούμε. Ο Μισελ Ντεντέ. Merci Madame Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες σας. Δεν σας κρύβω την ικανοποίησή μου γιατί βλέπω πως η οικονομία και οι φορείς του γεωργικού κόσμου αποτελούν εκ νέου την προτεραιότητα μιας προεδρίας. Νομίζουμε πως αυτό είναι καλό σημάδι, καλό ιονός. Πολύ δύσκολα ραντεβού σας περιμένουν. Σίγουρα θα έχετε ένα σημαντικό ραντεβού στον ΠΟΕ και ορισμένοι μάλιστα πιστεύουν ότι μέσα στους 5-6 μήνες που τους επόμενους θα μπορέσουμε επιτέλους να φτάσουμε σε μια συμφωνία στον γύρο της Ντόχα. Πώς σκοπεύετε να ε, ε, επιμείνετε στις προτεραιότητές μας τα θέματα που παραμένουν, δηλαδή φυτογενομικά, ε, ευημερία των ζώων ε, και ΚΟΑ, ε, που είναι πολύ σημαντικά στο δικό μας ευρωπαϊκό μοντέλο που θέλουμε εδώ να το περισπιστούμε στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Και τώρα, τελευταία από τις 17 παρεμβάσεις που έγιναν, κόρτες λάστρα. Señora Κυρία Υπουργέ Εσπινόσα, καλώς ήρθατε. Ευχαρίστηση είναι να είσαστε στην Ευρωβουλή για να μας ε, εξηγήσετε τις πρωτοβουλίες πολύ ορθές πιστεύω της Ισπανικής Προεδρίας για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη Πέθρου. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση θέλω να θέσω. Ποια είναι η άποψή σας, τι πιστεύετε ότι χρειάζεται η ΚΑΠ, ένα δίκτυο ασφάλειας όσον αφορά τις αγορές, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητή Ελένα, μετά από την ε, σωρία αυτών των ερωτήσεων, έχει όλο το χρόνο για να απαντήσεις. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για όσα θα μας πεις και για το τι θα καταπραίνεις τις ανησυχίες μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και θα προσφερθώ και για κάτι άλλο. Επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο, θα σας αποστείλω και γραπτές απαντήσεις, στον καθένα ξεχωριστά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά με σειρά παρέμβασης περίπου. ανάλογα με τα όσα ρωτήσατε. Στην κυρία Γκαρθία θα ήθελα να πω τα εξής. Μας ε, μίλησε για την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκο γενικά και μετά υπέβαλε ορισμένες ερωτήσεις και προτάσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής. Μιλάμε για την αναθεώρηση μιας συμφωνίας στον αγροτικό τομέα μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της Βαρκελόνης του 1995, όπου συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρου εμπορίου το 2010, τότε που θα τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Στο 2005 δόθηκε μία νέα όθηση στο όλο ζήτημα και τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή διαπραγμάτευσης με το Μαρόκο. Αυτά είναι τα συμφραζόμενα τα οποία γνωρίζουμε και γνωρίσαμε. Έκτοτε ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να σας πω ότι μετά από αίτημα διαφόρων χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, η εντολή ενήχε και μία ρήτρα σε σχέση με τα ευαίσθητα προϊόντα ως προς τις ε, εξαγωγές του Μαρόκου. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την παραγωγή της Ισπανίας με την παραγωγή του Μαρόκου. Θεωρούμε ευαίσθητα λοιπόν όλα τα πιο ευάλωτα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις και κλειδονισμοί της κοινωτικής αγοράς. Μία άλλη πτυχή που έπρεπε να λάβουμε υπόψη είναι η εξής. Όταν μιλάμε για τέτοιες συμφωνίες, πολλές φορές σκεφτόμαστε τι παράγουν τρίτες χώρες κάτι το οποίο μπαίνει στα κοινοτικά δεδομένα και ξεχνάμε ότι σε αυτές τις συμφωνίες και εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να εξάγουμε σε εκείνες τις χώρες. Κάτι το οποίο αφορά μεταποιημένα προϊόντα κυρίως που παράγονται στις μεσογειακές χώρες ανάλογα με το input που χρειαζόμαστε, ανάλογα με το input παραγωγής. Πολλές φορές μιλάμε για μεταποιημένα προϊόντα, για γεωργικά προϊόντα, για προϊόντα κτηνοτροφίας, μεταποιημένα, που μπορούν αφορούν, να αφορούν παραγωγή και ξέρετε ότι πολλές φορές ως προς όπορο και πευτικά υπάρχει μεγάλη κατανάλωση στο Μαρόκο. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι οι μηχανισμοί ελέγχου. Δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου. Όμως είναι περίπλοκοι και γι' αυτό πολλές φορές ε, υπάρχουν καθυστερήσεις ε, δεδομένων. που υποστηρίζουν αυτές τις συμφωνίες και δεν τα έχουμε σε πραγματικό χρόνο αυτά τα δεδομένα. Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση αυτή και εργάζεται εδώ και μερικούς μήνες έτσι ώστε να μας προσδώσει μηχανισμούς που να διευκολύνουν τον έλεγχο εισαγωγών-εξαγωγών υπ' αυτή την έννοια. Με αυτό το διτό χαρακτήρα δηλαδή. Ευρωπαϊκή Ένωση, Τρίτες Χώρες και Τούμπαλιν. Άρα το διάβημά σας, ε, το οποίο γνωρίζουμε, το οποίο ήδη γνωρίζαμε, ε, θα το αναλάβει και η Ισπανική Προεδρία και θα το αντιμετωπίσει το Ειδικό Συμβούλιο Γεωργίας. Και βεβαίως θα συναποφασίσει και το Κοινοβούλιο. Γιατί ε, οι προβλέψεις οι χρονικές μπορεί να υπερβούν την Ισπανική Προεδρία. Αλλά υπάρχει ένα ορισμένο χρονοδιάγραμμα. Αν μπορέσουμε να επιταχύνουμε τόσο το καλύτερο για να βελτιώσουμε τους ελέγχους στα πλαίσια της εκπεριτροπής Προεδρίας. Η κυρία Ερνάνς αναφέρθηκε στο έγγραφο που αφορά το μέλλον της ΚΑΠ. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ισπανική Προεδρία προσδίδει μεγάλη σημασία στο μέλλον της ΚΑΠ. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στα έγγραφα τα οποία καταρτίζουμε και, τις, και στις θέσεις του Συμβουλίου. Θα θέλαμε όμως να προωθήσουμε μια ανοιχτή συζήτηση, μια συζήτηση που να μας εμπλουτίσει που να μας δώσει όλα τα δεδομένα από τα κράτη-μέλη. Και αυτό περιλαμβάνει και άλλα θέματα που ανέφερε η κυρία Ερνάντεθ. Δεν θα θέλαμε να έχουμε ένα έγγραφο όπου, το οποίο δεν θα είναι απότοκο συζητήσεων. Θα δούμε και θέματα συγχρηματοδότησης καθώς και θέματα που αφορούν εξασφάλιση εισοδήματος. Η κυρία Ερνάντεθ γνωρίζει πολύ καλά τη θέση της Ισπανικής Προεδρίας. Εγώ δεν είμαι εδώ υπό την ιδιότητά μου ως Υπουργός Γεωργίας, αλλά ως υπεύθυνη της Προεδρίας. Η Ισπανία εδώ και 30 χρόνια προβάλλει ασφάλειες γεωργικού εισοδήματος που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο και αναγνωρίζονται και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες και αν θέλετε μπορούμε να, να τις θέσουμε σε διάθεση όλων των κρατών μελών όπως ε, κάναμε ορισμένες φορές για να ελέγξετε τη βιωσιμότητά τους και τη σκοπιμότητά τους για να προωθηθεί μια παράλληλη διάρθρωση σε όλα τα κράτη-μέλη ενδεχομένως. Αυτό θα ήταν ένα από τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης της αγοράς. Ίσως είναι σκόπιμο μέσο, υπάρχουν και άλλα και θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα το Φεβρουάριο στο Συμβουλίο Υπουργών Γεωργίας. Θα ήθελα όμως να επιμείνω ως προς το εξής. Ήδη από την δική μας Προεδρία θεωρούμε απαραίτητους, απαράβατους τους ε, μηχανισμούς αγοράς έναντι σεναρίων κλειδονισμών της αγοράς. Δηλαδή ως προς την ΚΑΠ πέρα του 2013. Εδώ ανοίγω μία γενική παρένθεση, έτσι ώστε όλοι να το σκεφτούμε από κοινού. Εδώ και τρία χρόνια Ε, ασχοληθήκαμε με θέματα που άπτονται κλιματικών αλλαγών, αντικσοτήτων του κλίματος και ούτω καθεξής. Γνωρίσαμε δηλαδή μία αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Αυτό δεν αφορούσε μόνο τις ζωοτροφές, αλλά όλα τα παράγωγα προϊόντα κτηνοτροφίας, αυξήθηκε η τιμή του ε, πετρελαίου, των λιπασμάτων, των σιτηρών στη διεθνή αγορά και γνωρίσαμε μία, μία ε, απαράμιλη ε, αύξηση τιμών των ζωοτροφών. Αυτό... Μέσα σε αυτό το σενάριο μια μεγάλη ανησυχία για τις επιπτώσεις ε, όσον αφορά τους ε, καταναλωτές ε, αυτό το κόστος των τροφίμων. Και είχαμε και άλλη ανησυχία, την σπανίδα δηλαδή συγκεκριμένων προϊόντων ακόμα και εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Ξαφνικά όλα αυτά εξομαλύνονται. Περνάμε όμως πάλι σε μια διεθνή παγκόσμια κρίση και τώρα η μεγάλη μας για το κύριο μέλημα μα είναι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να έχουν ένα δίκαιο εισόδημα που θα διασφαλίζουν. Ή με άλλα λόγια, κάθε ένα και όλοι οι κρίκοι τη αλυσίδα που συναποτελούν την αλυσίδα τη παραγωγή να έχουν ένα δίκαιο εισόδημα όσον αφορά τη δραστηριότητά του και την παραγωγή πρόσθετης αξίας, προστιθέμενη αξία. κάνουμε λόγο για το πρόσφατο παρελθόν και μιλάμε για δύο καταστάσεις που διαμετρικά είναι θα έλεγε κανείς διαφορετικές και αντίθετες. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε να συντεριάξουμε. Να μην πλήτεται η Ευρώπη από τέτοια δυσμενή φαινόμενα. Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα μας δίνει μια συγκεκριμένη σταθερότητα έναντι αυτού του ευμετάβλητου χαρακτήρα που έχει επιπτώσει σε όλους. Από το γεωργό στον κτηνοτρόφο, κάποιες φορές ε, θετικά αρνητικά και φυσικά πλήττει και έχει επιπτώσει στο τέλος τέλος και στον καταναλωτή, είτε θετικά είτε αρνητικά πάλι και στη συνέχεια θα, έχουμε ευκαιρία, θα έχω ευκαιρία να ε, παραμείνω και να σχολιάσω αυτά περισσότερο, ιστερότερα. Και το θέμα για το οποίο είναι λόγος από πλευρά Ερνάντεθ είναι για την πολιτική για τα δάση. <clears throat> Όπως επίσης είναι γνωστό και σε σχέση και με τοποθέτηση άλλων ευρωβουλευτών για να μην νομίσει κανείς ότι μονοπολώ τις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις σε σχέση με αυτή την παρέμβαση θα αναφερθώ και εκτενέστερα και στα άλλα στον κύριο Καπόλας ο οποίος έκανε λόγο τώρα για διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα για την απασχόληση μίλησε που και εγώ θα ήθελα να ε, σκεφτούμε κάτι που έχει γενικότερο χαρακτήρα ως σκέψη. Αν κάνουμε μια ανάλυση αυτών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των μηνών που ζήσαμε αυτή την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις που είχε αυτή η κρίση στον γεωργικό τομέα, στον κτηνοτροφικό τομέα. Πιθανώς τότε θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε, μία και σε όλα τα, σε κάθε ένα και σε όλα τα κράτη-μέλη <clears throat> είναι ε, εκείνος ο οποίος έχασε λιγότερες θέσεις απασχόλησης ή παγίωσε κιόλας ή και κάπως λίγο αύξησε την απασχόληση. Όμως αν δει κανεί ε, τον συσχετισμό σε σχέση με του ε, ανέργου ε, που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα, ίσω θα βρίσκαμε ένα μεγαλύτερο αριθμό. Αυτά τα δύο που σα είπα δεν είναι αντιφατικά. Αυτή τη στιγμή Στι περισσότερε περιπτώσει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο γεωργικό τομέα και ο κτηνοτροφικό τομέας έχει πλεονάσματα από άλλε βιομηχανικέ δραστηριότητε ή υπηρεσίε που είχαν μεγαλύτερη απώλεια δραστηριότητα και απορρέει ότι πρέπει να κάνουμε και αυτή την ανάλυση επίσης. Να δούμε ότι ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις υπάρχει ανταπόκριση καλύτερη και απάντηση καλύτερη από άλλοτε. Ας κάνουμε μια πρόσθετη προσπάθεια, ακόμα μια προσπάθεια, ώστε αυτή η απασχόληση να είναι σταθερή απασχόληση και να υλοποιεί και να ανταποκρίνεται στους άλλους στόχους που εμείς προσπαθήσαμε να ε, θεσπίσουμε και να επιτύχουμε. Και αυτονόητο και φυσικό είναι ότι όταν κάνουμε λόγο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε μόνο λόγο για το άθροισμα των 27 κρατών μελών ατομικά από πλευρά του. Η ΚΑΠ πρέπει να ε, ανταποκρίνεται και να λαμβάνει υπόψη τι ευαισθησίε όλων και κάθε ενό από τα κράτη-μέλη. Και αυτή η ΚΑΠ πρέπει πραγματικά να είναι δίκαια, να το πετύχουμε να είναι δίκαια. Και πρέπει να δίνει απαντήσει σε ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες των διαφορετικών κρατών. Επίσης, άλλος Ευρωβουλευτής στη συνέχεια εξέφρασε μια θέση και είπε ότι πρέπει, είπε, είναι ο κύριος Σικέρσκι, Σικερέσκι, αν δεν κάνω λάθος και προφέρω το όνομα σωστά, και είπε για την πολυμορφία της γεωργίας που υπάρχει και με διαφορετικά μεγέθη στα κράτη-μέλη. Όμως έχουμε και τον πλούτο που μας ε, συνεπιφέρει αυτή η γεωργία. Ο μεγάλος πλούτος της πολυμορφοποίησης και των διαφορών που υπάρχουν. Και αν θέλουμε η ΚΑΠ να είναι μια κοινή αγροτική πολιτική, τότε αυτή η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να δίνει απαντήσεις ή μέσω μιας αρχής επικουρικότητας με ένα περιθώριο ελιγμών για τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν ή με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά από μια ορεινή ορεινή ας πούμε γεωργία μέχρι και την γεωργία που δεν θα είναι ορεινή αλλά παιδινή. Και για χώρες που έχουν διαφορετικά κλιματολογικά χαρακτηριστικά και χώρες που έχουν πάλι τελείως διαφορετικά ε, στοιχεία όσον αφορά το κλίμα από άλλες. Ας δραχθούμε τις ευκαιρίες. Κάνουμε λόγο για την αγορά καταναλωτών, την ευρύτερη και μεγαλύτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε όλοι την ίδια ζήτηση τροφικών προϊόντων, δεν εκινούμε από την ίδια αφετηρία, δεν εκινούμε από τις ίδιες γαστρονομικές παραδόσεις. Αυτός είναι ο πλούτος μας όμως και ο πλούτος μας είναι επίσης αυτός που επιθυμούμε να δώσει απαντήσεις στην γεωργία της Ευρώπης με, παρα, με παραγωγές ε, διαφοροποιημένες και διαφορετικές μεταξύ τους. Παρόλες τις διαφορές θα πρέπει όμως να είναι δίκαια η αντιμετώπιση τους και εξισορροπημένη. Και έτσι θέλω να τοποθετηθώ στην παρέμβαση του κυρίου Καπόλας. Στη συνέχεια άλλος Ευρωβουλευτής ανέφερε το πόσο ευμετάβλητος είναι ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων πόσο εμβρευστό βρίσκεται και για την δραστηριότητα για παράδειγμα μεταξύ των κτηνοτρόφων που είναι από τις πιο ευαίσθητες γιατί από μια σειρά παραγωγών ολόκληρων που έχουν μια περίοδο ζωής, ένα κύκλο ζωής ευρύτερο στην περίπτωση του γάλακτος και όταν κάνουμε ε, λόγο για την νοπή κατανάλωση, κατανάλωση νοπού γάλακτος, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο πιο ευαίσθητος. Πρέπει εδώ μεγαλύτερη προσπάθεια να καταβληθεί όσον αφορά τους κτηνοτρόφους και για την παραγωγή. Απαιτούνται έλεγχοι ποιότητας και για την ασφάλεια της ε, διατροφής ε, ανώτατου επίπεδου, πολύ απαιτητική έλεγχη. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, τα ίδια τα ζώα, οι αγελάδες, για να μπορούν ε, να παράγουν αυτό το γάλα ως προϊόν, χρειάζονται πολλούς μήνες για να μπορούν να πετύχουν την οριμότητα εκείνη από πλευρά σώματος και ηλικία τους για να μπορούν να παράξουν αυτό το γάλα. Και πάλι εδώ έχουμε δύο άκρα που αντιμετωπίζουμε μεταξύ των δύο. Δεν είναι δυνατόν άμεσα να υπάρξει προσαρμογή ζήτησης και προσφοράς άμεσα. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό μέσα σε αυτές τις στενές περιόδους για την οριμότητα του ζώου. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ ευαίσθητος και τόσο πολύ περίπλοκο σύνθετος αυτός ο τομέας και τα προβλήματα και είναι ευμετάβλητο και ευαίσθητο όσον αφορά αλλαγές στη ζήτηση και την προσφορά και στις τιμέ. Αυτό οδήγησε από πλευρά των ομάδων υψηλών αξιωματούχων που αυτή τη στιγμή ε, μελετούν και αυτά τα θέματα και έχουν δρομολογηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό να είναι ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο θέμα για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το γάλα Υποβάλλονται λοιπόν τα αποτελέσματα αυτών των μελετών στα τελευταία Συμβούλια Υπουργών. Έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα για τη δική μας την Ισπανική Προεδρία και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις εκθέσεις και αυτές τις μελέτες που τώρα υπάρχει αρκετά μεγάλη περίοδο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέλιξη των αγορών. Οι συζητήσει, ε, ο προβληματισμό που έγινε από τι ομάδε υψηλών αξιωματούχων από την Επιτροπή για να αναζητηθούν αυτέ οι προοπτικέ μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και όπω εσείς ο ίδιο είπατε πρέπει να συναγάγουμε συμπεράσματα από αυτή την κρίση για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Επίση χρειάζονται και άλλα μέσα. Άλλα μέσα μόνο αυτά τα μέσα διαχείρισης της αγοράς ε, που για αυτά κάνω διαρκώς λόγο σε εσά εγώ πρέπει να υπάρξουν και άλλα. Να κάνω μια αναλογία εδώ. Θα είχαμε προτίμηση να υπάρξει και θα μια εξισορροπητική δραστηριότητα και εδώ αυτό μπορεί να θεωρηθεί εγχείρημα ακροβατικό. Όμως για να μπορέσει αυτό το θέαμα το οποίο συνεπάγεται συγκεκριμένους κινδύνους Πρέπει να υπάρξει και ένα δίκτυο ασφάλειας για αυτούς τους ακροβάτες ε, που θα περπατούν στο τεντωμένο σκηνή, ώστε αν υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα να μην χτυπήσουν και τραυματιστούν και ε, υπάρξει ε, πρόβλημα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και για το γεωργικό τομέα και για τον τομέα στην κτηνοτροφία. Να υπάρξει ένα δίκτυο ασφάλεια. Ένα δίκτυο ασφαλεία το οποίο έναντι οποιασδήποτε ανεξέλεγκτη κατάσταση θα ήταν αν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα, αυτό το δίκτυο ασφάλειας θα δρούσε και δεν θα υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις ούτε για την απασχόληση ούτε για την οικονομία γενικότερα. Και νομίζω τούτων λεχθέντων ότι κατάφερα να απαντήσω, απαντώ στις παρατηρήσεις ε, ε, συναδέλφου Ευρωβουλευτή που αναφέρθηκε στα θέματα των γαλακτοκομικών και θέματα αγοράς ε, και για αυτόν τον ρόλο που πρέπει να δώσουμε στη γεωργία μέσα σε ένα πλαίσιο ε, της σημερινής αγοράς. Επίσης, για την παρέμβαση σε σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το θέμα του ΠΟΕ, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, εγώ είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που λένε ότι πρέπει να συνάψουμε μια συμφωνία Ντόχα το δυνατόν γοργότερα. Αυτή η συμφωνία της Ντόχα και συμπίπτω και συμφωνώ με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν σε σχέση με τον Επίτροπο για τη γεωργία, πρέπει να μπορέσουμε να το κάνουμε με εκείνα τα οποία έχουμε ήδη επιτύχει σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική στο παρελθόν, με το κεκτημένο μας. Έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις, έχουμε τροποποιήσει σε βάθος πολύ σημαντικά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να επεξηγήσουμε καλά αυτές τις θέσεις, να τις προαπίσουμε θετικά και να τεθούν επιτραπέζεις ακριβώς αυτά τα οποία ε, έχουν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μιλήσουμε για τους βιομηχανικούς τομείς, ε, για παράδειγμα, και για τα θέματα που είναι τόσο σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επίσης και για άλλες δραστηριότητες, ώστε όλα αυτά να ευνοηθούν μέσα στην μεγάλη αυτή παγκόσμια αγορά, όπου θα ρυθμίζονται και θα διανοίγονται δυνατότητες. Η κυρία Γέκλε αναφέρθηκε στην παρέμβασή της στο ότι η ομάδα, η, η σχέση συνεργασίας που πρέπει να δημιουργηθεί, η ομάδα, το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία είναι απαραίτητο στοιχείο. Είχα την ευκαιρία να διαβάσω την παρέμβαση του Επιτρόπου που θα ήθελα να σας πω ότι συμμερίζομαι κατά 100% της θέσεις ε, και που αυτό το οποίο ε, εκτιμώ ότι μπορούμε να κάνουμε είναι σε αυτή την τριγωνική σχέση συνεργασίας να είμαστε το δυνατόν καλύτεροι στη συνεργασία μας για την προάσπιση των γεωργικών και αλλιευτικών συμφερόντων. Όμως έγινε λόγος και για τον ρόλο της γυναίκας στον χώρο της υπαίθρου επίσης. Τώρα εγώ πιθανώς εδώ σε σχέση με κάποια παρέμβαση που έγινε ίσως παρεμεινεύθηκε και σε σχέση με την τοποθέτηση του κυρίου Ανιώ θέλω να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα. Δεν πρόκειται εδώ για υποχρεωτικές διατάξεις και ρυθμίσεις που θα επιβληθούν σε κάποιους. Πρόκειται για ένα πεδίο ισότιμο για όλους που θα διασφαλίσουμε. Και όταν κάνουμε λόγο για ισότητα, χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά και επιτρέψτε μου να το κάνω αυτό προσωπικά το ότι η γυναίκα, λέω, στον χώρο της υπαίθρου υφίσταται διπλή αρνητική μεταχείριση. Πρώτον, επειδή είναι γυναίκα και δεύτερον επειδή ζει στον χώρο της υπαίθρου ως γυναίκα. Ας τερματίσουμε αυτή την κατάσταση. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Δεν πρέπει να κοστίζει χρήματα και να είναι δαπανηρό κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Ανιώ έκανε ένα σχόλιο και είπε οι γυναίκες και νομίζω αυτό λεξί μπορώ να το αναφέρω έτσι, εργάζονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ε, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ακόμα και οδηγούν, λέει, τρακτέρ. Και θέλω να πω και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των εκμεταλλεύσεων, η γυναίκα και ο άνδρας ή μόνο ο άνδρας. Ποιος είναι εκείνος που παίρνει τις ενισχύσεις ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΑΠ, η γυναίκα και ο άνδρας που εργάζονται κατά 50% εξίσου, δηλαδή εξημισίας ή ο άνδρας μόνο αυτό θέλω να σας διαβιβάσω ως μήνυμα. Πολλές φορές δεν κάνουμε λόγο για παραπάνω χρήματα ως κονδύλια. Το μόνο που θέλουμε είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες νομοθετικές να αναλυφθούν που θα αντανακλούν αυτή την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών που πιστεύω εγώ ότι είναι απόλυτα αναγκαία. Αλλά και πέρα από αυτό το πλαίσιο, αν κάποιο. και δεν θέλω να με παρεμηνεύσετε εδώ, να ε, παρανοηθεί αυτό, προσέξτε, αν κάποιο δεν το θεωρεί επαρκέ αυτό το θέμα της ισότητας, σκεφτείτε κάτι άλλο. Θέλουμε να έχουμε έναν χώρο τη υπαίθρου ζωντανό. Θέλουμε να, είμαστε, να πολυμορφοποιήσουμε τα πράγματα όπω αναφέρθηκε. Θέλουμε να διατηρήσουμε και να διασφαλίσουμε τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Ε, τότε δεν απομένει άλλο δρόμο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα και τι ικανότητες τη γυναίκα. Γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει οτιδήποτε άλλο. Και απλά και μόνο και βιολογικά Ας πάρουμε λοιπόν την λύση που ταιριάζει καλύτερα και είναι πιο σκόπιμη. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να εκφράσω αυτή την προσωπική άποψη για την ισότητα που μας αφορά όλους και που θα κάνει μια κοινωνία δικαιότερη, να είμαστε δικαιότεροι. Πράγμα που πρέπει να γίνει. Και αυτό το συνδέω, χωρίς να έχω αναφέρει το όνομα, με αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκαρθία Πέρες, που είπε ότι σε σχέση με αυτόν τον προβληματισμό, τον ευφυή προβληματισμό για την δυνατότητα να, έχουν, να εγκατασταθούν με διαρκή χαρακτήρα στον χώρο της υπαίθρου αυτοί οι άνθρωποι. Διότι σε σχέση και με τις ε, διεθνείς αγορές ε, και την, ε, τον ανταγωνισμό είναι αδιάφορη η ερώτηση ή ο, στόχος. Πρέπει να υπάρχει πρώτη ύλη. Αυτή η πρώτη ύλη παράγεται στον χώρο της υπαίθρου. Αλλά αυτή η πρώτη ύλη παράγεται χάρη σε χιλιάδες, μυριάδες γεωργούς και κτηνοτρόφους Ευρωπαίους που ζουν στην υπαίθρο και που στη συνέχεια περνάνε στις εθνικές αγορές, στα, ε, στις διεθνείς αγορές ή στις ε, βιομηχανίες ε, στα εργοστάσια μεταποίησης. Αν αυτοί οι άνθρωποι, οι γυναίκες και άνδρες δεν είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι στον χώρο της υπαίθρου, δεν θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους και να μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Με τον ίδιο τρόπο που δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά αν δεν είχαμε και νέους, νέους ανθρώπους. Αυτός ο συνδυασμός νέοι άνθρωποι και γυναίκες νομίζω για τους λόγους που τώρα δεν μπορούμε μπορούμε να συζητήσουμε εδώ. Έχουν, ε, έχουμε διαφορετικές σχέσεις και αναλογίες ισορροπίας με ξεχωριστά χαρακτηριστικά για τους νέους μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορέσαμε να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά για τις γυναίκες, αυτές τις δυνατότητες για τις γυναίκες. Ένα παράδειγμα για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπάθησε να έχει θετική μεταχείριση και αντιμετώπιση των γυναικών και είδε ότι κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο και δεν ήταν δυνατόν επειδή δεν υπήρχε αυτή η υποστήριξη από πλευρά κοινοτικών οδηγιών ή κανονισμών σε κοινοτικό επίπεδο. Μια άλλη από τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που παρουσιάστηκαν από τον κύριο Μαρτίνετ ήταν το θέμα των κονδυλίων από πλευράς προϋπολογισμού. Τι είναι εκείνο το οποίο σκεφτόμαστε εμείς ως Προεδρία. Εμείς ως Προεδρία θεωρούμε ότι σήμερα θα ήταν βιαστικό να κάνουμε λόγο για συγκεκριμένα ποσά ως κονδύλια. Δεν με ακούσατε να αναφέρω ένα συγκεκριμένο ποσό, έτσι δεν είναι. Έκανα λόγο για ένα υπαρκή προπολογισμό όσον αφορά τα κονδύλια. Γιατί, διότι λοιπόν, εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε κάθε μια και όλες τις κοινοτικέ πολιτικές με επαρκή τρόπο. Όταν θα έχουν σχεδιαστεί αυτές και κάθε μία από αυτέ ξεχωριστά, θα ξέρουμε ότι θα κοστίζουν χ ψ κονδύλια από πλευρά ευρώ. Και αυτό θα δώσει την δυνατότητα να διαμορφωθεί ο αναγκαίο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αντίθετα πούμε, έχω 100 και αρχίσουμε να κάνουμε παζαράκια ή αρχίζουμε να ε, μειώνουμε και στα μέσα του δρόμου δεν θα είχαμε χρήματα, θα είχαμε περικοπές ή μια, έναν, ένα συγκεκριμένο αριθμό προβλημάτων για την ανταπόκριση κονδυλίων και αναγκών. Σήμερα κάνουμε λόγο για τις ανάγκες που πρέπει να δούμε από πλευράς κονδυλίων και αυτές να μπορέσουν να διαμορφωθούν όταν θα έχουν αποσαφινιστεί οι ε, στόχοι και οι ανάγκες. Αυτό είναι κάπως αυτό το οποίο με άλλα λόγια εννοούσε ο κύριος Μαρτίνεθ, έτσι δεν είναι. Και πιστεύω ότι με τα θέματα αυτά έμεσα με την υποστήριξη για την ανάπτυξη που ανάφερε συγκεκριμένα για το θέμα του Μαρόκου π.χ. Πιστεύω ότι το γνωρίζουμε σαφώς αυτό και το έχουμε συνειδητοποιήσει. Φυσικά, ίδια η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στην βοήθεια που χορηγεί στην ανάπτυξη ανταποκρινόμενοι και στην δημιουργία πλούτου ως ανάγκη σε άλλες χώρες. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με έναν τρόπο συμβατό που να συνάδει με τους στόχους και τις ανάγκες της Ευρώπης. Και αυτό είναι μια πρόσθετη προσπάθεια. Αλλά πάλι και εδώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι η λιδία λήθος. Να είμαστε ικανοί να μπορέσουμε στις άλλες γενναίες να δώσουμε την ευκαιρία να μπορέσουν να ζήσουν στις τρίτες χώρες με καλύτερο τρόπο από ό,τι ζουν οι άνθρωποι εκεί σήμερα. Και εμείς δεν μπορούμε μπορούμε να ξεχνάμε ότι αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο σε όλη αυτή τη διαδρομή. Για τον κύριο Λεφόλ που έκανε λόγο για την περιβαλλοντική συνιστόσα, την περιβαλλοντική διάσταση. Λογικό, λογικά εγώ στην πρώτη μου παρέμβαση εκείνο που είπα είναι ότι πρέπει να διαμορφώσουμε μια γεωργική πολιτική και να την, της δώσουμε τέτοια χαρακτηριστικά, όχι μόνο με τα στοιχεία που είχε ιστορικά, όπως για παράδειγμα τα τρόφιμα, τα υγιή, καλά τρόφιμα και ποιότητας αναβαθμισμένα, αλλά η συνεισφορά που υπάρχει στο περιβάλλον να διατηρηθεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας ζωντανό αλλά επίσης και η συνεισφορά που κάνει η γεωργία και η κτηνοτροφία για ένα μέλλον που θα μπορεί να είναι καλύτερο όσον αφορά την θετική επιρροή για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Υπάρχει και μια άλλη σειρά θεμάτων που στη συνέχεια θα αναφερθώ σε αυτά πιο γενικά, διότι καλύφθηκαν σε πολλές από τις παρεμβάσεις σας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι της Ελλάδας εδώ, το ελληνικό πρόβλημα, που λογικό είναι ότι είναι ένα σημείο και εμεί ως Προεδρία το δεχόμαστε αυτό, ένα σημείο υπό τα διάφορα που θα πρέπει να εξεταστεί στο επόμενο ε, Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας για να το μελετήσουμε και να το εξετάσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να, επιλύσουμε, να αντιμετωπίσουμε και επιλύσουμε τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Όσον αφορά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από την κυρία Κανιέτε για την δίκαιη και ισομερή κατανομή και επιμερισμό, νομίζω απάντησα όταν απάντησα προηγούμενα κατά κάποιο τρόπο στον σύντροφο Καπόλας, Καπόλας Σάντος. Με τον ίδιο τρόπο, όπως δόθηκε απάντηση όσον αφορά την πολυμορφοποίηση και όσον αφορά και τις διαστάσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τα πολύμορφα στοιχεία. Ο κύριος Μπερλάτο αναφερόταν στην πολυλειτουργικότητα της γεωργίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ με, θα, αναφερθώ σε αυτό το σημείο. Η πολυλειτουργικότητα εντάχθηκε στις, ε, στην κοινή αγροτική πολιτική εδώ και κάποια χρόνια. Πρέπει να συνεχίσουμε να την ενδυναμώνουμε και να την ενισχύουμε γιατί αυτή, αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος που πρέπει να έχει και στο μέλλον ο χώρος της υπαίθρου. Αυτός ο κύκλος δηλαδή, ο κύκλος που πρέπει να εξετάζεται και να διαμορφώνεται ώστε ακριβώς ο χώρος της υπαίθρου να είναι ζωντανός, πλούσιος και όχι μόνο με χαρακτηριστικά μονοκαλλιέργειας πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού όσον αφορά τις δυνατότητες ε, του κόσμου που ζει στον χώρο της υπαίθρου. Θα προσπαθήσω λοιπόν τώρα να δώσω μια επεξήγηση ευρύτερη για θέματα που καλύφθηκαν από τον κύριο Κορτές μέχρι και πολλούς άλλους που παρενέβησαν πιο πριν και που αφορούν γενικότερα θέματα αλλά επίσης αναφέρονται στο να υπάρξει αυτή η δυνατότητα ένταξης ή πλαισίου πραγμάτων που πολλές φορές φαίνεται να μην είναι συνεκτικά και συμβατά που όμως δεν συμβαίνει αυτό. Κοινή αγροτική πολιτική. ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική. Πρέπει να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε αυτό το σενάριο πέρα από το ορόσημο του 2013, όπου η γεωργία και η κτηνοτροφία θα πρέπει να έχουν αυτόν τον προϋπολογισμό που θα είναι ισχυρός και συνεπής και συνεκτικός. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, όπω εκείνε τι προκλήσει που συνδέονται με τι κλιματικέ αλλαγέ ή τις, ε, ε, το περιβάλλον ή τη βιοπικιλότητα ή την ενίσχυση και τη βοήθεια στην ανάπτυξη ή που ε, θα σχετίζονται με την υλοποίηση των στόχων τη χιλιετία. Και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο ιστορική σημασία έργο και πρόκληση τη διατροφική ασφάλεια, ασφάλεια των τροφέμων και διασφαλισμένη σύντηση από πλευρά προϊόντων για όλου. Αυτό γίνεται λοιπόν Λοιπόν μέσα στο πλαίσιο του χώρου της υπέθρου. Στο χώρο της Υπέτρου, σαν συνέπεια, πρέπει να έχουμε όχι μόνο τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά επίσης την πολυλειτουργικότητα, ώστε ο κόσμος να αισθάνεται άνετα, να μπορεί να ζει ευχάριστα εκεί και να συνεχίσει να ζει στο χώρο της Υπέτρου. Μέσα όμως σε αυτόν τον κόσμο που μου κάνουμε λόγο γενικά για αυτόν, έχουμε τη γυναίκα ξεχωριστά Πρέπει να εξισώσουμε αυτή τη γυναίκα, να της δώσουμε προϋποθέσεις να είναι ίση. Για αυτή την πρώτη ύλη που παράγεται στον χώρο της υπαίθρου από πλευράς ε, γεωργίας και κτηνοτροφίας. Πολλές φορές πάει στη μεταποιητική βιομηχανία και στα εργοστάσια, όχι μόνο ως ένα πρωτογενές προϊόν μεταποιητική βιομηχανία που και εδώ και πάλι πρωτοπόρος είναι παγκόσμια και που θέλουμε και επιθυμούμε να μπορέσει να προσαρμοστεί όχι μόνο στους στόχους και προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να μπορεί να συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος παγκόσμια στην αναδιαμόρφωση της συμφωνίας και στρατηγικής της Λισαβόνας που την αποκαλούμε στρατηγική 2020 και που πρέπει να έχει και να δίνει το καλύτερο σενάριο και τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα από πλευράς μας. Ανταγωνιστικότητα που επιπλέον την αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας να εμπλουτίσουμε όσο γίνεται με ομάδες υψηλού επίπεδου που αναπτύσσουν το έργο τους αυτές τις στιγμές και να συμπληρωθούν με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν όσον αφορά νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια ανάπτυξης υπαίθρου. Και σαν συνέπεια όλων αυτών, μέσα σε αυτό το μεγάλο ιστό για να μπορέσουν όλα αυτά να λειτουργήσουν και για την μεταπητική βιομηχανία και όλα τα άλλα, χρειαζόμαστε αυτό το δίκαιο ασφάλειας που σας είπα για τη διαχείριση των αγορών το οποίο θα το συζητήσουμε στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2010 και που θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις στις κρίσεις συγκυριακές ή δομικές που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις κρίσεις τιμών ή και στην ε, ε, διάθεση ε, γεωργικών προϊόντων και στον ευμετάβλητο χαρακτήρα των αγορών και στα προβλήματα της αλυσίδας της διατροφής των τροφίμων. Αυτό το σενάριο θα είχε τον καταναλωτή τώρα που πρέπει να καλύψουμε. Πώς σκεφτόμαστε και τι έχουμε υπόψη να κάνουμε ως Ισπανική Προεδρία. Τι μπορεί να γίνει για να λειτουργήσουν όλα αυτά και τι, τι μπορεί να γίνει. Να βελτιωθεί αυτή η αλυσίδα ώστε κάθε ένας από τους κρίκους και όλοι οι κρίκοι να ενισχυθούν. Πέρα από αυτό ως εκκίνηση η συζήτηση μπορεί να πάει και πιο πέρα, πιο μακριά σε σχέση με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Και πρέπει ίσως να συνενώσουμε το καλύτερο θα ήταν αυτό προσπάθειες και αρμοδιότητες και ικανότητες. Αλλά και αυτό πάλι είναι μια πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σας ενθαρρύνω και σας προτρέπω να ανοίξετε αυτή την προοπτική να γίνει αυτό. Διότι εκεί μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις που μπορούν να βρεθούν και να δοθούν που σήμερα δεν τις έχουμε ακόμη. Κάποιες από αυτές ε, όσον αφορά την ε, παρουσίαση, την διοργάνωση της ενιαίας ρύθμισης αγορών και άλλες που πρέπει να έχουμε ανοιχτό ορίζοντα και μεγαλόπνοο σχεδιασμό για να βρούμε τις σωστές απαντήσεις. Νομίζω έφτασα στα όρια τα χρονικά που είχαν τεθεί, έτσι δεν είναι. Τώρα, θέλω να ολοκληρώσω προσπαθώντας να μπορέσω να ανταποκριθώ, να απαντήσω σε εκείνα τα θέματα πιο εξειδικευμένα που δεν ήταν δυνατό να το, υπάρξει άλλη τοποθέτηση λόγω έλλειψης χρόνου. Θα το κάνω αυτό σε σχέση με κάθε έναν από αυτά ξεχωριστά. Και τώρα ένας τελευταίος προβληματισμός για κάτι που θυμήθηκα, για κάτι το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν, όταν έγινε λόγος ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι μια δαπανηρή, λέει, ακριβή πολιτική. Εδώ θα πρέπει επίσης να μας προβληματίσει και κάτι άλλο και να το σκεφτούμε και αυτό. Ας βγούμε από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ας δούμε τι κάνουν οι ΙΠΑ, οι Αμερικάνοι και ας κάνουμε μια απλή σύγκριση στοιχείων μεταξύ των ΙΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> έχει πάνω πάνω την διαφάνεια και ας κάνουμε και μια δεύτερη σκέψη ως προβληματισμό για κάτι που είναι πιο κοντά σε μας. Τι γίνεται σε σχέση με την ε, ε, ε, Ελβετία και να πάμε και ως την Ιαπωνία που σχεδιάζει μια πολιτική γεωργική κατά και παρόμοια με εκείνη της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έκανα λόγο για χώρες που εξετάζουν ξεχωριστά τα δικά τους θέματα. Είπα, η Ιαπωνία, <clears throat> ε, την ε, Ελβετία μπορούμε να προσθέσουμε κι αλλά μην ξεχάσουμε αυτά κάνουμε λόγο για θέματα που όλοι γνωρίζουμε κάνουμε λόγο για κάτι που σε καμιά χώρα προηγμένη χώρα δεν έχει απεμποληθεί ο στόχος. Δηλαδή για τη διατροφική ασφάλεια, την επισητιστική ασφάλεια. Εδώ δεν κάνουμε λόγο για μια χώρα μόνο, κάνουμε χώρο για 27 χώρες που έχουν συνενωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι αξιόλογο και πρέπει να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτή την περηφάνεια που είναι περηφάνεια ευρωπαϊκή, να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές και περιβαλλοντικά να είναι πιο αηφόρα η παραγωγή, η ευρωπαϊκή παραγωγή. Εδώ ακριβώς βρίσκονται τα κέντρα στα οποία θα εργαστούμε ως Ισπανική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητή Ελένα Εσπινόζα. Πραγματική ακρόαση περάσατε σήμερα. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που μας δώσατε και είμαι βέβαιος και πεπισμένος ότι στο Ισπανικό εξάμεινο θα έχουμε μια σημαντική περίοδο εντατική συνεργασίας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ένα λεπτό διάλειμμα. Σιωσιγή ήθελε να πήγε να πει ο πρόεδρος, εννοούσε διάλειμμα.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

Συνεχίζουμε τις εργασίες μας με την παρουσίαση μελέτης σχετικά με τον καπνό. Δίνω το λόγο στον κύριο Ούντο Κένλε που είναι ο συγγραφέας της μελέτης. Χαιρετίζω και τους εκπροσώπους της Επιτροπής υπενθυμίζω στον κύριο Κάινλε ότι έχει 15 λεπτά για την παρουσίασή του και στη συνέχεια θα γίνει μια συζήτηση, γρήγορη συζήτηση, γιατί έχουμε και ένα άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη σε σχέση δηλαδή με τις περιοχές με μειονεκτήματα και την ειδική έκθεση της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω κι εγώ Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω. Έχω κάνει μια μελέτη για τον καπνό. Το ξέρω πως ο καπνός είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Από τη μια πλευρά υπάρχουν καπνοπαραγωγοί, από την άλλη υπάρχουν το θέμα της δημόσιας υγείας και οι οργανώσεις καταναλωτών που δεν θέλουν να προωθείται ο καπνός και τα προϊόντα του. Η ομάδα μελέτη που δεν ήταν μόνο καθημαϊκή ή οικονομολόγοι, παραγωγή, ήταν και εκπρόσωποι τη γεωρική ανάπτυξη από την Ισπανία. Είχαμε μισό χρόνο περίπου, έξι μήνες περίπου να κάνουμε αυτή τη μελέτη και η βάση της μελέτης αυτής ήταν διάφορα έγγραφα της Κομισιόν των ε, Εποπτών καθώς και η διαφοροποίηση του καπνού, όπου το δικό μας τμήμα ήταν ο συντονιστής και είχαμε και μία συνάντηση μετά ως οργανώσεις των καπνοπαραγωγών, αφού είχαμε κάνει το πρώτο σχέδιο της μελέτης μας. Τα σημεία κλειδιά για τον καπνό είναι τα εξή. Καταρχήν ξεκινήσε με την ανακοίνωση του Προέδρου Πρόντι πως ο καπνός είναι μια μη βιώσιμη καλλιέργεια και ότι σιγά σιγά θα πρέπει να καταργηθεί η καλλιέργειά του. Μετά από αυτό ακολούθησε η απόφαση σχετική του Συμβουλίου και ξεκίνησε μια πολιτική για το πώς θα γίνει αυτό και φέτος φτάσαμε στη δεύτερη φάση που σημαίνει ότι το 50% των επιδοτήσεων ε, ε, σταματούν και από την επόμενη χρονιά γίνεται η διαφοροποίηση και η μεταρρύθμιση του τομέα. Είναι δύσκολο να γίνει η διαφοροποίηση του καπνού, της καλλιέργειας καπνού, γιατί ο τομέας αυτός συνήθως αποτελείται από μικρές εκμεταλλεύσεις. Και αυτό για ιστορικούς λόγους, διότι σε πολλές περιοχές όπου καλλιεργεί το καπνός, Ήδη πριν από 50 χρόνια υπήρχαν αυτές οι καλλιέργειες και αυτές οι καλλιέργειες έδιναν ανέκαθεν δουλειά στην οικογένεια. Το 95% λοιπόν των εκμεταλλεύσεων καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούνται από λιγότερο από 15 εκτάρια. Κυρίως 5 είναι τα εκτάρια. Και η μόνο, ο μόνος πόρος εισοδήματος είναι η γεωργία για τις ε, οικογένειες αυτές. Άρα λοιπόν η διαφοροποίηση μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρχει μια πολύ ε, κερδοφόρα καλλιέργεια. Διαφορετικά οι εκμεταλλεύσει αυτέ θα ε, καταρρεύσουν. Ένα άλλο στοιχείο είναι το φύλλο. Ε, Προηγουμένω μιλήσαμε για την συμμετοχή των γυναικών στη Γεωργία. Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ο τομέα του καπνού είναι ο μόνο γεωργικό τομέα όπου έχουμε πολύ ψηλότερη ιδιοκτησία των εκμεταλλεύσεων από γυναίκες, από ότι οποιοδήποτε άλλος τομέας. Συνήθως βρίσκεται στο 10% πάνω από τον μέσο όρο των υπόλοιπων γεωρικών τομέων. Έπειτα υπάρχει επίσης το πρόβλημα πως η απασχόληση επίσης, οι θέσεις εργασίας καλύπτονται από γυναίκες. Είτε μόνιμη απασχόληση είτε εποχιακή απασχόληση λέμε. Είναι γυναίκες αυτές που δουλεύουν στα καπνά. Και κυρίως οι αυτές οι εκμεταλλεύσεις των γυναικών είναι εξαιρετικά μικρές. Όταν λοιπόν μιλάμε και λέμε ότι οι περισσότερες θέσεις είναι απαραίτητες για γυναίκες, είναι ηρωνικό. Είναι παράδοξο το να καταστρέφουμε αυτό το τομέα. Όταν άρχισε να σχεδιάζει την πολιτική αυτή η Κομισιόν, υπήρξαν δύο μικρές λεπτομέρειες που τελικά είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Η πιο εκτεταμένη αξιολόγηση επιπτώσεων έγινε από την Κομισιόν με αντικατάσταση του καπνού από σκληρό Τα αποτελέσματα δεν ήταν σωστά, γιατί οι γεωργοί συνήθως δεν κοιτάνε μόνο την κερδοφορία, αλλά το γενικό ε, εισόδημα, δηλαδή το ε, ακαθάριστο περιθώριο που είχαν ο καπνός έδινε πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Επίσης, υπήρχε ένας κανονισμός στο παρελθόν μέσω του οποίου η Κομισιόν έκανε διάφορες μελέτες για τον καπνό και για εναλλακτικέ λύσεις για τον καπνό. Όταν όμως σχεδίασαν τη μεταρρύθμιση, τα ταμεία πήγαν από μια κεντρική προσέγγιση της Κομισιόν στις εθνικές κυβερνήσεις, τα κονδύλια δηλαδή. Έτσι η Κομισιόν έχασε τον έλεγχο της ίδιας της πολιτικής. Μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις έδιναν χρήματα για αυτού του είδους τα προγράμματα διαφοροποίησης. Και αυτή ήταν και η αχίλιος πτέρνα του προγράμματος. Διαφοροποίηση τώρα, λέμε. Υπάρχουν 81.000, σχεδόν 82.000 ε, ε, εκμεταλλεύσεις, καπνοκαλλιέργειες. Το 95% πρέπει να κλείσει γιατί δεν παίρνουν χρήματα από επιδοτήσεις, επιβιώνουν ως καλλιέργειες μόνο όταν παίρνουν επιδοτήσεις. Αν αυτό συμβεί, αν αυτό γίνει θα χαθούν 250.000 με 280.000 θέσεις απασχόλησης στο γεωρικό τομέα δεν έχουμε πολύ και σε όλες τις χώρες, αλλά κύριε χώρε είναι αυτή τη στιγμή η Ιταλία, η Πολωνία και η Ισπανία και μετά η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Βουλγαρία μάλλον, που, που είναι σημαντική χώρα που καλλιεργείται ο καπνός. Έγιναν τέσσερις μελέτες για να ελεγχθούν οι δυνατότητε διαφοροποίησης. Η μία ήταν μία το πρόγραμμα Άστρα που το πλήρωσε τον Λεωνάρντο Νταβίντσι και εξέταζε την απασχόληση των απασχολούμενων αυτή τη στιγμή σε καπνοκαλλιέργειες. Τι θα γίνονταν όλοι αυτοί. Μια άλλη μελέτη έγινε από το Ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας και έπειτα ένα project για μελέτη της διαφοροποίησης και βεβαίως πρόσφατα μία έκθεση της ε, Κοσέγκα ε, για την ε, αξιολόγηση της μεταρρύθμισης. Συμπεραίνουν όλες αυτές οι μελέτες ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση στο καπνοκαλλιέργεια. Ποιο είναι το μέγεθος της ε, διαφοροποίησης. Όταν βλέπει κανείς μια εκμετάλλευση, βλέπει πως υπάρχουν εκμεταλλεύσεις μόνο ενός εκταρίου που καλλιεργούν κάθε χρόνο ε, καπνό. 12.500 ευρώ έχει εισόδημα. Συνήθως φυτεύουν ένα εκτάριο καπνό, έχουν παρόμοιο εισόδημα και παραδίπλα υπάρχουν άλλες εκμεταλλεύσεις. Αν θέλουμε να έχουμε εναλλακτικέ, θα πρέπει να φτάσουν σε ένα επίπεδο εισοδήματος περίπου 12.000 ευρώ. Γιατί διαφορετικά με λιγότερα χρήματα δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιταλία, ας πούμε, υπάρχουν πολύ καλές στατιστικές για ε, τον γεωργικό τομέα και συγκρίναμε τι λένε οι Ιταλικές στατιστικές για τα μοντέλα δηλαδή γεωργίας διάφορες καλλιέργειες ή κτηνοτροφία ή πτηνοτροφία. Αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι από τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων και τα χαρακτηριστικά τους ότι περισσότερες εκμεταλλεύσεις προχωρούν με ένα σχέδιο διαφοροποίησης των καλλιεργιών. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις χρειάζονται πολύ ψηλά ε, εισοδήματα για να μπορούν να διατηρήσουν ε, προσωπικό στις εκμεταλλεύσεις τους. Ποιε είναι οι πραγματικές ε, εναλλακτικές. Υπάρχουν αρωματικά φυτά, ενεργειακά φυτά, αγροτουρισμός, νέες καλλιέργειες ή συνέχιση της καλλιέργειας του καπνού αυτό που μπορούμε να δηλώσουμε είναι οι δραστηριότητες σε τέτοιες εκμεταλλεύσεις είναι αδύνατες. Γιατί ταυτόχρονα οι περισσότερες περιφέρειες ε, που καλλιεργούνται τα καπνά ήδη είχαν μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Χωρίς να λάβουμε υπόψη την ε, κρίση που διανύουμε την οικονομική. Όταν κάναμε λοιπόν την έρευνα είχαμε ερωτηματολόγια από 22.000 εκμεταλλεύσει. Μόνο πέντε από αυτές μπορούσαν να επιβιώσουν με καλλιέργειες ενεργειακών φυτών. Τα αρωματικά φυτά είναι πολύ δύσκολη η καλλιεργιά τους. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει μεγάλη συμβατότητα ε, προέρχονται από πολύ λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και υπάρχουν πολύ λίγες δυνατότητες για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καλλιέργειες και ο αριθμός των νεκταρίων είναι πολύ περιορισμένος. Τώρα, για μια μικρή εκμετάλλευση είναι απαραίτητο να έχει καλλιέργεια μεγάλης προστιθέμενης αξίας ή να είναι μόνο πρόσθετο το εισόδημα που περιμένει κανείς από αυτή την εκμετάλλευση. Με τους ε, γεωργούς των 5 εκταρίων δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορεί να φτιάξεις, ναι, να φτιάξεις ας πούμε να βάλεις εκεί πουλερικά. Αλλά αυτό που είδαμε πριν από δύο χρόνια με την μεγάλη αύξηση του κόστου των ζωοτροφών, αν δεν έχει κανεί επαρκή γη στην εκμετάλλευσή του, ώστε να φτιάχνει μόνο του τα σπόρια που ταζει τα ε, πουλερικά, οποτεδήποτε γίνεται μια τέτοια αύξηση κόστου, σταματάει και η παραγωγή. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη, δεν υπάρχει εύκολη λύση. Για τι μεγάλε εκμεταλλεύσει, ναι, αυτό είναι δυνατόν. Αλλά στον καπνό είναι πολύ λίγε οι μεγάλε εκμεταλλεύσει. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έκανε μια καλή μελέτη που μελέτησε το μέλλον των αγορών για τα φρούτα και λαχανικά Ιδιαίτερα στις περιοχές όπου καλλιεργείται ο καπνός υπάρχει ήδη μεγάλο επίπεδο, ψηλό επίπεδο παραγωγής φρούτων και λαχανικών. Όλες αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν όταν θα αρχίσει η ελεύθερη εισαγωγή από τις τρίτες χώρες και όταν συγκρίνουμε τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων, δείτε, δείτε στην Ελλάδα, στη Μακεδονία ας πούμε, εκεί υπάρχουν 7.000 εκμεταλλεύσεις για χανικά και φρούτα. Να βάλουμε κι άλλες 60 και άλλε 60.000 εκμεταλλεύσει, ε, θα καταστραφεί η αγορά όλων των άλλων περιοχών. Γιατί οι τιμές θα πέσουν και οι γεωργοί θα μείνουν ε, χωρίς δουλειά. Άρα δεν υπάρχει καμία λύση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Εδώ έχετε μία συνολική εικόνα ως προς τις ε, δυνατότητες. Εδώ βλέπετε πόσες εκμεταλλεύσεις υπάρχουν σε κάθε κατηγορία και βλέπετε ε, ότι κάτω από 50 εκτάρια έχουμε 22.000 εκμεταλλεύσεις. Άρα είναι ο τομέας που διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο. Τι γίνεται τώρα με τη μεταρρύθμιση για τον καπνό από το 2004. Μία συνέπεια όπως φαίνεται από τη μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν το 2003 και ήταν αναμενόμενο, ήταν ε, ότι κατά τη στιγμή της μεταρρύθμισης οι τιμές ανέβηκαν. Αυτό συνέβη σε ένα βαθμό. Και εδώ είδαμε ότι εξαντλήθηκαν τα αποθέματα. Βλέπετε λοιπόν ότι ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα 4% πολύ χαμηλό αριθμό παραγωγής αλλά το 1 ή 2% λιγότερο, λιγότερη παραγωγή μεταξύ του 2004 και του 2004 οδήγησε στην εξάντληση αποθεμάτων και τα μειούμενα αποθέματα οδήγησαν στην αύξηση των τιμών του καπνού. Όταν συγκρίνουμε λοιπόν τις τιμές από το 2007 η ΕΠΑ, ΕΕ, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες βλέπουμε ότι φτάνουμε τα 2 ευρώ ανά κιλό στη Βερόνα αλλά στην Ισπανία καταβάλλονται 50 cents ανά κιλό. Δηλαδή η τιμή του Μαλάου και της Βραζιλίας. What is clear is that the prices are going up. Άρα οι τιμές ακολουθούν ανωδική πορεία και ίσως αυξηθούν και μακροχρόνια. Θα υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν να φτάσουμε σε δίκαιες τιμές για τους καπνοπαραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορέσουν να καλλιεργούν χωρίς επιδοτήσεις. Άρα μπορούμε να διαιρέσουμε τις περιφέρειες σε τρία τμήματα. Υπάρχουν ορισμένες περιφέρειες ή χώρες όπου η αύξηση φαίνεται και ήταν και πολύ υψηλή. Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ρουμανία, στην Ελλάδα μόνο τα ανατολικά καπνά και Ιταλία. Αλλά στην Πορτογαλία δεν υπήρξε αύξηση, ούτε στην Ισπανία. Και υπάρχουν και περιφέρειες τώρα όπου έχει σταματήσει η καπνοκαλλιέργεια. Εδώ έχουμε και καλλιέργεια Βιρτζίνια, όπου το 50% και στην Ελλάδα το 50% των ανατολικών καπνών ε, σταμάτησε και στην Ιταλία σταμάτησε ολοσχερός. Αυτό σημαίνει, για να το ποσοστοποιήσουμε, έχουμε 11.000 εκμεταλλεύσεις όπου θα πρέπει να έχουμε διαφορετική δραστηριότητα, μετατροπή δραστηριότητα, αν πρόκειται να παραμείνουν ε, στην ε, παραγωγή και έχουμε 79.000 εκμεταλλεύσεις που μπορούν να κρατήσουν την κάπνο καλλιέργεια και να φτάσουν σε μια δίκαιη τιμή της αγοράς. Άρα προτείνουμε το εξής είτε στην πρώτη φάση που ήταν 100% καταβολή που θα πρέπει να παραταθεί αυτό σημαίνει αλλαγή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ' αυτή την έννοια και οι εκμεταλλεύσεις να παραμείνουν στην παραγωγή, στην καλλιέργεια είτε να έχουμε ένα ελβετικό μοντέλο όπου ορισμένοι φόροι μπαίνουν σε εθνικά ταμεία και έτσι οι καπνοκαλλιεργητές μπορούν να λαμβάνουν χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έναν πρόχειρο υπολογισμό για τις πληρωμές, αλλά πρόκειται για πολιτική απόφαση. Τώρα, για τις εκμεταλλεύσεις που θα πρέπει να στραφούν σε εναλλακτικέ δραστηριότητες ε, εδώ θα τα τελευταία δέκα χρόνια να προωθηθεί μια νέα καλλιέργεια. Έτσι ώστε να υπάρχει μια εναλλακτική καλλιέργεια μπορούμε να προτείνουμε μια καλλιέργεια που είναι πολύ καλή για το διαβήτη, δεν παράγει τοξίνες και αυτή η καλλιέργεια δεν χρειάζεται πολλές ε, επενδύσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο εξοπλισμό. Οι κλιματικές συνθήκες είναι οι ίδιες και δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές για τους ε, αγρότες, για τους καλλιεργητές. Τώρα βλέπουμε ποιες, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες της αγοράς. Βλέπετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 55 δις ε, αναψυκτικά, τα οποία καταναλώνουμε κάθε χρόνο. Άρα το, άμα το 10% ε, δοθεί για αυτή τη δραστηριότητα θα έχουμε 40.000 με συγχωρείτε εκτάρια δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η χρήση σαν προσθετικό τροφίμων, αλλά θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε ένα νέο προϊόν. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η σκοπιμότητα, να γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας για 10 χρόνια λοιπόν. Προωθήσαμε αυτό το project, να δούμε τη μηχανιστική δηλαδή της καλλιέργειας αυτής και μετά είχαμε μία αύξηση για το Ταμείο Καπνών για να δούμε κατά πόσο υπάρχει σκοπιμότητα. Επίσης και στο Βένετο και στη Γρανάδα στην Ισπανία έγινε αυτή η μελέτη που ήταν επιτυχής. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι στις ε, ε, χώρες αυτές, συν Βουλγαρία και Ρουμανία, αυτή η καλλιέργεια είναι α, εναλλακτική πραγματικά. Τον Οκτώβριο του 2009 ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας για να γίνουν δοκιμές για να δούμε σε ποιες εκμεταλλεύσεις μπορεί να προωθηθεί αυτή η εναλλακτική καλλιέργεια. Θα ήθελα να σας δώσω ένα σαφές παράδειγμα. Γιατί ως προς την διαφοροποίηση καλλιέργειας θα πρέπει να δούμε ποιες ήταν οι εξελίξεις. Το project αυτό το είχαμε προτείνει το 2005 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Είχαμε μία αξιολόγηση αλλά η Κομισιόν δεν είχε τα κατάλληλα κονδύλια. Άρα ήμασταν, υπολοιπόμασταν κατά πολύ. Άρα θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι νέες δυνατότητες. Κατά από αυτές τις συνθήκες ήταν αδύνατο να καλλιεργήσουμε το οτιδήποτε. Η Κομισιόν δεν μπορεί να προωθήσει τα προγράμματα έρευνας. Και ένα άλλο παράδειγμα με το, ε, το 2007 προτείναμε ένα άλλο project, αλλά δεν είχαμε καλή αξιολόγηση. Όμως αυτοί που αξιολόγησαν μας είπαν ότι το project αυτό δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί διότι αντικαθιστά τα καπνά. Δηλαδή στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας ακολουθήθηκε μια άλλη πολιτική ως προς τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Είναι δύσκολο λοιπόν να ε, φτάσουμε σε δύο διαφορετικές καλλιέργειες. Συμπεράσματα. Υπάρχουν εναλλακτικές, εναλλακτικές καλλιέργειες και τις βλέπετε στην έρευνα. Αλλά υπάρχει περιορισμός ε, σημασίας. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει επίπτωση σε πολλές εκμεταλλεύσεις. Για τις μικρές εκμεταλλεύσεις το καλύτερο θα ήταν να έχουμε οποροφόρα. Αλλά υπάρχει απειλή, η εξής απειλή, να μην έχουμε ανοιχτές αγορές οι καλές τιμές. Αυτό αφορά και τις υδατοκαλλιέργειες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νέες καλλιέργειες. Σήμερα δεν υπάρχει καμία εναλλακτική που να είναι έτοιμη προς εφαρμογή. Μία άλλη έκβαση γίνεται λόγος για τον δεύτερο πυλώνα, αλλά στον δεύτερο πυλώνα δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα. Επίσης δεν υπάρχουν μέτρα για έρευνα. Άρα όταν μιλάμε για διαφοροποίηση καλλιέργειας, ε, αυτό είναι κάτι που χρήζει περαιτέρω ε, έρευνας. Η Γενική Διεύθυνση Άγκρη θα πρέπει να ασχοληθεί με διαφοροποίηση καλλιεργειών και να φτάσουμε σε μια νέα χρηματοδότηση καπνών για να προτείνουμε εναλλακτικέ ε, καλλιέργειες όπως αυτή τη στέβια ρεμπαουντιάνα. Εάν λοιπόν γίνει χρηματοδότηση θα πρέπει να δούμε και πόσες ε, θέσεις θα απολεστούν, θέσεις εργασίας. Πού θα προωθηθούν αυτές οι εναλλακτικές καλλιέργειες και το, ο δεύτερος πυλώνας γιατί η καπνοκαλλιέργεια μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτές τις απώλειες, να τις αντικαταστήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι έρευνες διαφοροποιημένων καλλιεργιών. Στη ΣΥΠΑ έγινε αυτή η μεταρρύθμιση στον τομέα του καπνού πολλά χρόνια πριν και φέτος έληξε αυτή η μεταρρύθμιση. Χρειάζονται όμως 10 χρόνια επιπλέον έτσι ώστε να προωθηθούν εναλλακτικέ καλλιέργειες και να υπάρξει νέος προσανατολισμός για τις εγκαταλεύσεις και το ίδιο θα γίνει εδώ. Χρειαζόμαστε ακόμα 10 χρόνια και μετά από μεγάλες και επίπονες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Mulțumesc, domnule pentru σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας ε, υποβάλω μία ερώτηση εγώ ως προς το νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υπάρχουν δύο αντιφατικά ζητήματα επιτρέπουμε ή δεν επιτρέπουμε την στέβα για ανθρώπινη κατανάλωση. Και, για τον... και μάλλον ο κύριος Σμίθ έχει το λόγο για να υποβάλει ερώτηση. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίζω και ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο ήταν μια ένεση αδρεναλίνης που μας έκανε η έκθεση του και πραγματικά ε, σας ε, ευχαριστώ, ειλικρινά σας ευχαριστώ για τη μελέτη που κάνατε. Είναι κάτι που αξίζει να το εξετάσουμε. Εγώ βέβαια διαφωνώ ε, κάθετα με τα δικά σας πορίσματα που λέτε στη σελίδα 113 ε, που λέει ότι με την υπόθεση της συνέχισης της καταβολής των επιδοτήσεων και αν αυτό καταστεί από πολιτική άποψη εγώ πραγματικά διαφωνώ με αυτή την υπόθεση και θα το συζητήσουμε και δεν είμαστε κατά της επιδότησης, δεν είμαστε κατά της επιδότησης ευάλωτων περιοχών ή οικονομικά ευαίσθητων περιοχών ή τα διάφορα προγράμματα για γεωργία και περιβάλλον κτλ. Και υπάρχουν άλλα προγράμματα τα οποία ευχαρίστως εξετάζω. Υπάρχει, δεν υπάρχει φυσικά πρόβλημα με την ιδέα ότι ο καπνός δεν έχει καμία διατροφική αξία. Εντάξει, άλλα γεωργικά προϊόντα επίσης ε, δεν έχουν ε, τροφικά ωφέλη. Ο καπνός όμως είναι πολύ διαφορετικό προϊόν και οι επιπτώσεις δημόσιας υγείας ε, είναι πολύ σημαντικές και επηρεάζουν την οικονομία των χωρών μας και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό το προϊόν λοιπόν είναι αντικειμενικά διαφορετικό. Καταλαβαίνω πως υπάρχει εδώ ε, μεγάλος διχασμός για το θέμα, αλλά η δική μου ψηφοφόρη είναι ομόφωνη για αυτό το θέμα. Εμείς υποστηρίζουμε τις ευάλωτες δραστηριότητε και τις οικονομικά ευαίσθητες περιοχές, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο. Και δεν είμαι κανένα στρατευμένος ή ιστερικός. Αν ο κόσμος θέλει να καπνίζει, εντάξει. Αν θέλουν να καλλιεργούν καπνό, επίση α του αφήσουμε. Αν και αν μπορούν να κερδίζουν και λεφτά με αυτή την καλλιέργεια, εντάξει, τόσο το καλύτερο. Αλλά πραγματικά είμαι αντίθετο στη χρήση δημόσιου χρήματο όταν ε, φαίνεται σαφέ ε, πω οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι η μέτοχη των ε, εταιριών των καπνοβιομηχανιών. οι 250 με 280.000 εργαζόμενοι, οι 80.000 ίσως να είναι μόνιμα απασχολούμενοι, οι υπόλοιποι είναι εποχιακοί εργαζόμενοι και θα μπορούσαν ίσως να βρουν άλλες οικονομικέ δραστηριότητε. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ και όπως σας είπα, μα άναψε τα αίματα. Ε, διαφωνώ με τα δικά σα συμπεράσματα, αλλά είμαι ευχαριστημένος που φέρατε αυτή την μελέτη. Εγώ είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για κατασπατάληση δημοσίου χρήματο και δυσφημεί την ΚΑΠ. Θα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία αυτή της έκθεση για να εξακολουθήσω να υποστηρίζω την κατάργηση των επιδοτήσεων ε, του καπνού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κίνλι για αυτή την ενδιαφέρουσα ε, έκθεση που μας έκανε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι μόλις γίνεται λόγος για τον τομέα του καπνού θα πρέπει να υπογραμμίσουμε διάφορες επιτυχίες κλειδιά και η πρώτη είναι αυτό που ακούσαμε μόλις ότι δηλαδή είναι σημαντικό να μην βάζουμε αυτομάτως ένα ίσον ανάμεσα στην παραγωγή του καπνού και την καταπολέμηση του καπνίσματος στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι έχει προτεραιότητα η υγεία των Ευρωπαίων, αλλά ως εκπρόσωποι όλων των πολιτών είναι που επίσης σημαντικό να μην γνωρούμε τα προβλήματα ορισμένων πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών καπνού. Εγώ λοιπόν επιμένω για την μαζική απώλεια θέσεων απασχόλησης που θα είναι μια συνέπεια της μεταρρύθμισης στο τομέα και αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης, πράγμα το οποίο ε, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Για την άποψή μου λοιπόν πρόκειται για ένα κομβικό σημείο, το να θέσουμε δηλαδή στην καρδιά κάθε συζήτηση που αφορά το τομέα την ε, απασχόληση. Να σας θυμίζω ότι στην, για, τη χώρα μου, τη Βουλγαρία, υπάρχουν περίπου 37.000 οικογένειες που δουλεύουν σε αυτό το τομέα και η χώρα μας είναι η μεγαλύτερη δηλαδή καπνοπαραγωγός χώρα στην Ευρώπη και πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν κάνει παρά μόνο αυτό όλο τους ζωή. Κάθε λοιπόν προπαγγελματική ε, μετατροπή είναι ε, λεπτό θέμα. 50% από αυτούς είναι ε, ηλικία 40 με 60 και επιπλέον ο κατακαιρματισμός των γεών δεν διευκολύνει τα πράγματα και... Ε, υπάρχει και μια πτυχή που ήδη έχει τονιστεί, δηλαδή η θέση των γυναικών στον τομέα αυτό και στη Βουλγαρία είναι ένα πρόβλημα ανησυχητικό αυτό. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την πιο οικονομική πτυχή. Υπάρχει η κοινωνική απασχόληση, αλλά και η οικονομική πτυχή και εσείς αναφερθήκατε σε αυτό. Είναι ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες των περιοχών όπου καλλιεργείται ο καπνός. Στη Βουλγαρία είναι περιφερειακές περιοχές, οικονομικά μειονεκτικές και ε, γι' αυτό νομίζω ότι από τη στιγμή που προσπαθούμε να προτείνουμε λύσεις εναλλακτικέ, είναι σημαντικό να έχουμε ένα τακτικό διάλογο με τις εθνικέ κυβερνήσει για να προτείνουμε ακριβώ ε, μέτρα τα οποία να αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες ε, του τομέα και των περιοχών. Να κλείσω λέγοντα ότι ίσως η πάυση των επιδοτήσεων να είναι μια λύση επικριτέα, όμως ε, το να πούμε πως δεν υπάρχει άλλη λύση ή το να προτείνουμε εναλλακτικέ που το βλέπουμε με τη μελέτη δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικότητες του τομέα νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σταθούμε στα εξή, να βάλουμε την απασχόληση στην καρδιά των μελλοντικών μεταρρυθμίσεων και εν πάση περιπτώσει στη συζήτηση που αφορούν τη μεταρρύθμιση και την ευελιξία στην εφαρμογή που κατά την άποψή μου ε, δύο κριτήρια που θα μας επιτρέψουν να απαντήσουμε ίσως καλύτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, καθημερινά η παραγωγή. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για τα εξαιρετικά γαλλικά σας και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπεριλάτο. Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει τόσες σχολικές εκδρομές κάθε χρόνο όπου ερωτώμεθα πολλά και διάφορα. Μεταξύ των διαφόρων ερωτήσεων που μας υποβάλλονται είναι η εξής. Τι σημαίνει... Τι σημαίνει μορία, τι σημαίνει βλακεία. Η καλλιέργεια είναι ένα παράδειγμα μορίας. Τα διάφορα θεσμικά όργανα χρηματοδοτούν μελέτες σαν αυτές, σαν αυτή, για να δείξουν, την να δείξουν την βλακεία, τη μορία, διότι όλα καταδεικνύουν ότι το να θέλουμε να απαγορεύσουμε, να απαλείψουμε την καπνοκαλλιέργεια στην Ευρώπη είναι κάτι που δεν είναι καθόλου λογικό. Μα αυτό δεν είναι παραγελίο. Είναι γελίο, υπάρχουν διάφορα συμφέροντα που υπερασπιζόμαστε. Μιλάμε για κατάργηση του τομέα καπνοκαλλιέργειας μιλώντας για, με υγιεινίστικα κριτήρια. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί δημοσίως την καπνοπαραγωγή τη στιγμή που θα πρέπει να καταβάλει πολλούς πόρους για να θεραπεύσει αυτούς που καπνίζουν, τους καπνιστές οι οποίοι παθαίνουν καρκίνο. Βλακία, μεγάλη βλακία, διότι η Ευρώπη εισάγει το 75% των αναγκών της σε καπνά από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Πολλοί από τους εκλογείς του συναδέλφου που προανέφερε το γεγονός ότι αντιτίθενται στην ε, παραγωγή η καλλιέργεια καπνού είναι καπνιστές καπνίζουν αριμανίως και θα πάθουν καρκίνο του πνεύμονα. Λέει ο μιλητής, τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε, να εξασφαλίσουμε την υγεία του καταναλωτή ή να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να οδηγηθούμε στον όλεφρο χρησιμοποιώντας την καπνοκαλλιέργεια και καπνοπαραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι πεθαίνουν πολλοί γιατί για την παραγωγή καπνού χρησιμοποιούνται και καρκινογόνες ουσίες σε χώρες εκτός Ευρώπης. Εγώ δεν είμαι καπνιστής. Είχα τρεις συγγενείς που πέθαναν από καρκίνο του πνεύμονα. Ακριβώς επειδή κάπνιζαν. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα υπάρχουν εκείνοι που χρησιμοποιούν μια υγιεινίστικη λογική για να θέσουν σε κίνδυνο 500.000 θέσεις στην Ευρώπη χωρίς να δώσουν σοβαρές εναλλακτικές εναλλακτικές λύσεις ως προς την απασχόληση αυτών των παραγωγών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή τη μελέτη μας ε, εξέθεσε, μας έδωσε δεδομένα και δεν γνωμοδότησε. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές στην καπνοκαλλιέργεια. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν οικονομικές συνέπειες, ολέθριες συνέπειες, διότι οι καπνοκαλλιεργητές μας ε, εξασφαλίζουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα. Είδαμε την απασχολησιμότητα, μας μίλησε και η Ισπανίδα Υπουργός, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι γίνεται και με την γυναική απασχολησιμότητα. Αντί να ψάχνουμε άλλες θέσεις εργασίας, α κρατήσουμε αυτές που υπάρχουν και για τις γυναίκες, χωρίς να δημιουργούμε περισσότερη ανεργία. Με εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ανησυχούν ιδιαίτερα με τις τάσεις ανεργίας, τόσο που δημιουργούν περισσότερη ανεργία. Τώρα, ως προς τις περιβαλλοντικές σκέψεις επειδή μιλάμε για εγκατάλειψη της καλλιέργειας και επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικέ, φτάνουμε σε μια απερίμωση που γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι. Μιλάμε για την ΚΑΠ, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η καταπολέμηση κλιματικών αλλαγών αποτελεί κύριο γνώμονα το, της συλλογιστικής μας, ενώ σοβαρές μελέτες, σοβαρές μελέτες καταδεικνύουν ότι αυτό το θέμα των κλιματικών αλλαγών δεν έχει αποδειχθεί. Δηλαδή δεν είναι ένα ανθρωπογενές φαινόμενο. Άρα κατασπαταλούμε πολλούς πόρους, και τελειώνω πρόεδρε, για να καταπολεμήσουμε κάτι του οποίου τις ρίζες δεν γνωρίζουμε. Και αυτό πάμε ε, στην Κοπενχάγη όπου γνωρίζουμε τον κόλαφο των άλλων χωρών. Εάν λοιπόν θέλουμε να φτάσουμε σε μια διαφοροποίηση καλλιέργειας, ως προς την καπνοκαλλιέργεια. Θα πρέπει να δώσουμε χρόνο σε αυτό το τομέα να βρει εναλλακτικέ καλλιέργειες και να προωθήσει και την απασχόληση, να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Μπορούμε να ε, διαφοροποιήσουμε αυτό το τομέα, να τον αναδιορθώσουμε, αλλά ίσως αυτό μην είναι πάντα δυνατόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. εδώ και τέσσερις φορές μιλήσαμε για την διατήρηση της επιδότησης των καπνών, γιατί εδώ μιλάμε για οργική παραγωγή, καθαρά, πέρα από το θέμα του καπνίσματος και της καταχρήσης σε αυτό το τομέα. Ελπίζω για μία φορά οι γραφειοκράτες της ε, Κομισιόν να τα καταφέρουν. Ελπίζω να μην εθελοτυφλούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε ιδέες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε δύο εκθέσεις ακόμα που πρέπει να, να μας απασχολήσουν. Ο κύριος Παπαστάμκος. Το μικρόφωνο σας κύριε Παπαστάμκο. Μικρόφωνο. Παρακολουθήσω τη συζήτηση με επίκεντρο την υγεία, το δημόσιο αγαθό της υγείας ε, γιατί ε, η συζήτηση θα πήγαινε εις μάκρος και δεν είμαι και ειδικό. δηλώνω καπνιστής και υπήρξα και μέλος μιας οικογένειας καπνοπαραγωγικής στα παιδικά μου χρόνια. Αλλά αν ανοίγαμε το φάκελο δημόσια υγεία, τότε θα έπρεπε να φέρουμε πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα και κτηνοτροφικά στο τραπέζι των συζητήσεών μας. Δεν διερωτώ αν το ορμονούχο ο κρέας είναι περισσότερο ή λιγότερο επιβλαβές. Διαρωτώ με επίσης γιατί να υπάρχουν ποσοστώσεις στην εισαγωγή βοήου κρέατος από την Αργεντινή και να μην αφαιθούν τελείως ελεύθερες εισαγωγές βοήου κρέατος από την Αργεντινή. Μ' αρέσει περισσότερο το αργεντινό στέικ από ότι το, το εγγλέζικο. Γιατί, επομένως, εάν θέλουμε να πούμε κάτι, μην οχυρωνόμαστε πίσω από τη δημόσια υγεία που πράγματι συντρέχει στη συζήτηση την οποία συζητούμε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, πολύ απλά θέλω να πω το εξή. Δεν μιλούμε για τον καπνό, την καλλιέργεια καπνού ως μια βιώσιμη καλλιέργεια που να πάρει σε βάθος χρόνου. Δεν συζητούμε γι' αυτό. Μιλούμε για την μετάβαση. Για τη διαφοροποίηση. Αυτό είναι το, ήταν το ζητούμενο της μελέτης του Policy ε, Department για διαρθρωτικές και πολιτικέ και πολιτικέ συνοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να ευχαριστήσω από καρδία του συντελεστέ αυτή τη μελέτη. Μην μα διαφεύγει αυτό. Πώ θα διαφοροποιήσουμε την καλλιέργεια. Και κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε προοφθαλμών ημιορεινές περιοχές, μικρές, πολύ μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ένα χέκταρ, ένα εκτάριο, και πώς θα πείσουμε ανθρώπους τη ηλικία των 55 ετών, όπως είπε η κυρία Νεντέλτσεβα, των 60, των 50 και άνω, να μεταβούν σε ένα, στην καλλιέργεια άλλων προϊόντων. Περί αυτού μιλούμε. Δεν είμαστε εδώ ε, για να κάνουμε... Δεν είμαστε Επιτροπή Υγείας. Εγώ θέλω να σου πω ότι πράγματι στη χώρα μου, και τελειώνω με αυτό, ο αριθμός παραγωγών μειώθηκε, κάπλων παραγωγών, κατά 63% το 2004, η έκταση κατά 62% έχει μειωθεί και η παραγωγή μειώθηκε κατά 80%. Από 48.000 περίπου καπνοπαραγωγούς, οικογένειες, σήμερα μιλούμε για 14.500-15.000 οικογένειες. Αλλά πρέπει να έχω ως εκπρόσωπός τους μία πιστική απάντηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για σένα που ζει σε μία περιοχή που ο καπνός για σένα έχει οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, δεν μιλούμε για περιφέρειες, μιλούμε για τοπικές κοινωνίες, για, τοπικές, για μικρές περιοχές, πρέπει να, δώσω, να στείλω ένα μήνυμα ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση σου δείχνουμε έναν άλλο δρόμο. Περί αυτού νομίζω η συζήτηση την οποία διεξάγουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ πολύ. κύριε Πρόεδρε. Θέλω εκ προημίου να πω ότι δεν καπνίζω. Κάποτε στα νιάτα μου κάπνιζα. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω στον συνάδελφο, τον συνάδελφο Μπερλάτο να τον υποστηρίξω στην παρέμβασή του σε σχέση με την καλλιέργεια καπνού στην Ευρώπη. Ακόμα και αν τίποτα δεν κάνουμε και εγκαταλειφθεί, θα υπάρχουν καπνιστές στην Ευρώπη. Εγώ προτιμώ να έχουμε καπνό για τους καπνιστές στην Ευρώπη και να τον παράγουμε στην Ευρώπη αντί να τον εισάγουμε από αλλού. Και δεν το θεωρώ σκόπιμο εδώ να κάνουμε σταυροφορία κατά της καπνοκαλλιέργειας, της καλλιέργειας καπνού στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι ακόμα και με τις ε, ε, ε, τους τίτλους στα πακέτα σιγαρέτων είναι θανα, θανατηφόρο το κάπνισμα δεν τρόμαξαν οι καπνιστές συνεχίζουν να καπνίζουν δεν ήταν αποτρεπτικό αυτό και ένα άλλο παράδειγμα επί χρόνια οι ομάδες προστασίας ε, ζώων είχαν παρέμβει λέγοντας ότι παράλληλα με τις μεταφορές ζώων στον Λίβανο ότι αυτές είναι ανεδαφικές και δεν πρέπει να υποστηρίζονται ε, και πρέπει να είμαστε κατά του ότι τέτοια ζώντα ζώα θα μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα αυτά τα ζώντα ζώα έρχονται από την Αυστραλία, Νότια Αμερική στο Λίβανο. Έτσι μεταφέρονται εκεί. Και δεν ακούω τίποτα από τις ομάδες προστασίας ε, των ζώων πλέον. Έχει καθησυχάσει πλέον η συνείδηση των Ευρωπαίων. Και διαρωτώ με κατά πόσον είναι αξιόπιστοι κάποιοι που παρεβαίνουν με αυτόν τον τρόπο και πόσο αξιόπιστες είναι κάποιες τοποθετήσεις αυτού του είδους. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μία οδό, έναν τρόπο η δυνατότητα αυτή καλλιέργεια καπνού στην Ευρώπη σε εκείνες τις περιφέρειες όπου υπάρχει να μπορέσει να διατηρηθεί αλλά και να παρακαλέσουμε να ζητήσουμε από τους επιστήμονες και εδώ έχουν γίνει και προτάσεις τα επόμενα χρόνια να αναζητηθούν σκόπιμες εναλλακτικές καλλιέργειες που μπορούν να εξευρεθούν ώστε εκείνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να βρουν μια τέτοια εναλλακτική καλλιέργεια να μπορέσουν να διασφαλίσουν την ύπαρξή τους στον χώρο της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βοητσαϊκόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα υποστηρίζω τον κύριο Ντάσκε, και τον κύριο Μπερλάτο. Και Ευχαριστώ εκείνους που είναι υπεύθυνοι για αυτή την έκθεση που νομίζω μας βοήθησαν και μας βοήθησε αυτή η έκθεση και στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο και όπως είπε ο κύριος Μπερλάτο μπορέσαμε να επανέλθουμε σε αυτό το ε, θέμα αρκετές φορές κατά το αμέσο παρελθόν. Υποστηρίζω το θέμα αυτών των ε, ενισχύσεων. Δεν είναι δυνατόν ε, να μπορέσει ο τομέας της καπνοκαλλιέργειας διαφορετικά να είναι βιώσιμος και να μπορεί να διασφαλιστεί η ύπαρξή του. Αν δει κανεί τώρα τα ναρκωτικά, τις ναρκωτικές ουσίες ε, και αν υπάρχει απαγόρευση, τότε αυτό είναι σαφές ότι έχει επιπτώσεις όμως εδώ κάνουμε λόγο για την καλλιέργεια καπνού που είναι νόμιμη και όπου η διανομή και η κατανάλωση καπνικών προϊόντων είναι νόμιμες υποθέσεις. Δεν είναι ένα παράνομο ε, είδος ουσίας ναρκωτικών και είναι ένα παράδειγμα αυτό το ότι ακολουθεί η κοινότητα την οδό της ελάχιστης αντίστασης. Και εδώ κατηγορούμε δηλαδή στο τέλος τέλος τα ίδια τα θύματα εκείνο το οποίο κάνω είναι δεν μπορώ να δεχθώ ε, τέτοιου είδου επιχειρήματα. Δεν κάνουμε λόγο για τις μεγάλες εταιρείες καπνοπαραγωγών ε, και εδώ μιλάμε για μικροκαλλιεργητές. Δεν είναι μεγάλης έκτασης καλλιέργειας. Πολλές φορές είναι πολύ μικρής έκτασης καλλιέργειας, οικογενειακές καλλιέργειες κιόλα. και που μόνο το οικογενειακό ε, εισόδημα μπορούν να διασφαλίσουν το πολύ πολύ. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα όταν συζητάμε για άλλου είδους ε, ε, δράσεις και δραστηριότητες. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, κάνουμε λόγο για πολύ μικρής κλίμακας, μικρής έκτασης καλλιέργειας, πολύ μικρής έκτασης. Πρέπει να υπάρξει κάποια ελάχιστη κατανόηση κάπως και να υπάρξει και πολιτική βούληση. Φυσικά υπάρχει μια συνιστόσα υγείας όσον αφορά θέματα υγειονομικά εδώ, αλλά δεν είναι δυνατό να ισοπεδώσουμε τους μικρούς καλλιεργητές και καλλιεργητές και να πούμε έτσι θα επιλύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία. Mulțumesc. Τέσσερις ακόμα ζητάνε το λόγο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είσαστε σύντομοι, διαφορετικά θα είναι αδύνατον να ασχοληθούμε με τις δύο άλλες εκθέσεις που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, διότι έχουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα να υποβάλουμε τροπολογίες. Ο κύριος Σιεκέρσκι έχει το λόγο.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 Ξέρουμε ότι η παραγωγή του καπνού δεν έχει σχέση με το πόσο καπνίζει ο κόσμος. Έτως ή άλλως έχουμε πολύ ποιοτική παραγωγή στην Ευρώπη. Ε, τα καπνά που παράγουμε είναι πολύ ποιοτικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι δεν θέλουν να υποστηρίξουν αυτές τις παραγωγές. Ε, είναι παράλογη αυτή η στάση. Σας ευχαριστώ κύριε Χόσλινγκ. Μόνο πολύ σύντομα. Όταν τίθεται το ερώτημα αν πρόκειται σε σχέση με τον αριθμό αυτό, αριθμό θέσεων πλήρου απασχόληση ή δευτερογενού απασχόληση, για να έχουμε ρεαλιστικά αριθμητικά στοιχεία, θεωρώ υπερβολικό αυτό τον αριθμό που αναφέρθηκε ω θέσει πλήρου απασχόληση. Υπερβολικό αριθμό. Και σε σχέση με το, αυτό το οποίο αμφισβητείται περισσότερο σε σχέση με την γεωργική πολιτική είναι η ασυνέπεια τη πολιτική μα που αποφασίζει να κάνει κάτι κατά της ε, κατάχρησης των καπνικών προϊόντων και μετά τίθεται το ερώτημα ναι ενισχύουμε την καλλιέργεια καπνού την ενισχύαμε με μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτή είναι μια πολιτική που είναι ασυνεπής και παντού να λέει κανείς ότι καλύτερα να έρχεται από την Ευρώπη να προέρχεται αυτός ο καπνός και αν είναι βλαπτικός ας έρχεται από τα δικά μας χωράφια και όχι από ξένα ε, δεν είναι επιχείρημα αυτό ε, και τουλάχιστον και σε σχέση με τα ναρκωτικά να πει κανείς ε, να, έρχεται, να έρχονται αυτά από την Ευρώπη για να τα ελέγχουμε καλύτερα δεν είναι επιχείρηματα αυτά. Κυρία Κλάς, τελευταία ομιλήτρια αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και δυνατότητες και ξέρω ότι από τη δική μου περιφέρεια που υπάρχουν λίγοι ε, καπνοκαλλιεργητές όμως παραπονούνται ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα λένε να διασφαλίσετε μια μεγαλύτερη προθεσμία ως διορία για να υπάρξουν εναλλακτικέ λύσεις. αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το θέμα όμως είναι ότι οι νέες εναλλακτικέ καλλιέργειες ε, μπορούν να επιτραπούν, έχουν αδειοδοτηθεί στην Ευρώπη. Πόσο θα διαρκέσει το θέμα της αδειοδότησης και πόσο σε σχέση με τις ε, αποκλειστικέ τέτοιε ε, καλλιέργειες ή φυτίες μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τους καπνοκαλλιεργητές. Διότι μπορεί να υπάρχει και ευρύτερο ενδιαφέρον. Τουλάχιστον για τους καπνοκαλλιεργητές θα πρέπει να στοχεύουμε αυτό να μπορέσει να ισχύσει. Ε, κύριε Κίνλε, θα ήθελα να απαντήσετε, αλλά σε δύο λεπτά αν γίνεται. Λοιπόν εντάξει, στα γερμανικά μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι έχουμε μελετήσει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες ως πρόπτικη και η αλήθεια είναι δεν υπάρχουν τέτοιες πολλές. Γενικά ο κύριος Σμίθ έχει δίκιο ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε, έχουμε καθήκον να υποστηρίξουμε. Όμως πρέπει να δούμε και τα στοιχεία ως facts, ως γεγονότα και το γεγονός αν πάτε και επισκεφτείτε αυτές τις ε, περιοχές ε, καπνοκαλλιέργειας ε, δεν υπάρχουν και πολλά άλλα που να μπορεί κανείς να κάνει και το θέμα των θέσεων απασχόλησης στη μελέτη εξειδικευμένα αναφέρονται τα θέματα των θέσεων απασχόλησης είναι περιορισμένη απασχόληση θέσει εργασία. Είναι σαφέ αυτό, απόλυτα σαφέ. Όμω, αν δείτε τι περιφέρειε αυτέ, δεν είμαι ε, επιστήμονας αλλά είμαι ο ίδιος ε, και είχα, έχω εργαστεί σε, σε τέτοια εκμετάλλευση ε, τότε οι χρονικές περίοδοι σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο εργάζεται κάποιος σε κάποια καλλιέργεια και στην επόμενη περίοδο, στον επόμενο κύκλο με, με άλλη καλλιέργεια αλλού ή εναλλάξ και έτσι κατά τη διάρκεια ολόκληρου έτους διασφαλίζουν το εισόδημά τους οι γεωργοί αυτό κάνουν εναλλακτικά. Αυτό το οποίο σχεδόν αποκλείεται είναι αυτός ο μεγάλος αριθμός ε, γεωργών που επικεντρώνονται σε λίγες περιφέρειες πραγματικά να μπορέσουν να βρουν μια διαρκή θέση απασχόληση αλλού. Αυτό το θεωρώ ότι, θεωρώ ότι αποκλείεται. Δεν είναι δυνατόν. Και για αυτόν τον λόγο, και μόνο και για αυτόν τον λόγο, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν είμαι ε, φίλο ε, των μεγάλων καπνοβιομηχανιών εγώ ίδιος κάπνιζα, σταμάτησα όμως εδώ και χρόνια να είμαι καπνιστής πια. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι μόνο για αυτόν τον λόγο προτείνεται και προτάθηκε τα μέτρα αυτά να αλλάξουν, να τροποποιηθούν, να προσαρμοστούν ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη χρονική περίοδος για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Δύο φορές ε, ε, έγινε λόγο ε, για αυτές τις καλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αδειοδότηση, αλλά υπάρχει ευκαιρία να γίνει αυτό, διότι αν είχε γίνει το θέμα, είχε ολοκληρωθεί το θέμα της αδειοδότηση, θα γινόταν αυτό το οποίο είπε ο Ευρωβουλευτή. Και για να υπάρξει ειδικά κάτι υπέρ των καπνοκαλλιεργητών και των συνεταιριστών καπνοκαλλιεργητών, θέσαμε από την 1η Οκτωβρίου 2009 αυτή την ε, πρωτοβουλία όπου συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση κάνουμε λόγο για 7 συνεταιρισμούς ε, που περίπου 10.000 ε, εκτάρια καλλιεργούνται εκεί όπου αυτή η εναλλακτική δυνατότητα πρέπει να αναπτυχθεί από πλευράς τους. Και για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα που προβλέπεται ε, εξειδικευμένα σε ένα τομέα να παραμείνει ανοιχτός και να μείνει ανοιχτός για τους καπνοκαλλιεργητές να μπορέσουν εναλλακτικά να δραστηριοποιηθούν εκεί. Αυτό έχει προβλεφθεί. Σας ευχαριστώ. Πολύ λυπάμαι, σας ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είχατε και πολύ χρόνο να μας απαντήσετε. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Προχωράμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση για τη γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα για τον ειδικό έλεγχο υγείας. Το 54% της επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται, ε, θεωρείται ότι αφορά περιοχές με μειονεκτήματα. Και προτείνουμε ευελιξία. Από την άλλη προβλέπετε ότι θα πρέπει στα κράτη-μέλη Ο κύριος Χόφμαν εκπροσωπεί την Κομισιόν. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, πρόκειται για μια έκθεση που αφορά στο χρονικό διάστημα μετά το 2013. Θα πρέπει λοιπόν αυτά όλα να τα λάβουμε υπόψη μας πριν τεθούν σε ισχύ. Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε ήδη ότι περίπου το 35% της καλλιεργούμενης γης είναι τα, οι περιοχές που είναι ε, σε μειονεκτική θέση και για τέτοιου είδους περιοχές μιλάμε. Δεν μιλάμε ούτε για ορεινές περιοχές, ούτε για άλλες περιοχές, παρά μόνο για τις μειονεκτούσες. Αυτές λοιπόν οι περιοχές αυτή τη στιγμή ορίζονται από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πάνω από 100 κριτήρια που ορίζονται από τα κράτη-μέλη και αυτός ε, είναι ο λόγος ε, που το ελεγκτικό συνέδριο έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το θέμα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια που δημιουργούν ανισορροπίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη και είναι επίσης γεγονός ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα το οποίο οδηγεί σε αυτόν τον διαχωρισμό είναι πολύ διαφορετικό και αντιμετωπίζεται τελείω διαφορετικά στα 27 κράτη-μέλη. Η Κομισιόν προσπάθησε να βρει καινούργια κριτήρια και προτείνει τώρα οκτώ νέα κριτήρια τα οποία μπορώ να σας τα αναφέρω ε, όπως είναι η δομή, οι ε, ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις ρίζες και επίσης και η μορφή της κλητίος. Και με βάση αυτά λοιπόν τα κριτήρια και ε, με βάση τις νέες οριακές τιμές θα υπάρξει νέος διαχωρισμός των περιοχών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, όπως σας είπα για την ε, αντισταθμιστική εισφορά. Εκείνο που έχει επίσημα σημασία είναι κατά πόσον η γεωργική πολιτική ή η αντισταθμιστική εισφορά ε, προάγει ε, σωστά τις, τις σωστές εισφορές ή όχι. Στην πρόταση της Κομισιόν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνδυασμός ανάμεσα σε αυτά τα κριτήρια, δεν υπάρχει και δυνατότητα συνδυασμού υπάρχει ε, μια ε, τιμή εισόδου της τάξης του 66%. Ε, Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεσή μας αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα απλή, γιατί κανονικά θα έπρεπε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στα κράτη-μέλη οποτεδήποτε εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια. Και θα ήθελα να σας πω ότι η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη αυτά τα ε, νέα κριτήρια ε, να τα προσωμιωθούν ε, στις, στις νέες περιοχές. Βεβαίως οι κάρτες αυτές μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν παρότι από ορισμένα κράτη-μέλη αναφέρεται ότι έχει γίνει αυτή η προσωμείωση. Φαίνεται λοιπόν από μία ε, πρώτη αξιολόγηση των δεδομένων ότι αυτά τα κριτήρια δεν λειτουργούν παντού και θα υπάρξουν μικρές ή μεγάλες μετατοπίσεις. Στην έκθεση λοιπόν κατόπιν τούτου προτείνεται ή συστήνεται αν θέλετε ότι είναι απολύτως απαραίτητο ε, να δούμε εμείς αυτή την προσωμείωση πριν τελικά καταλήξουμε σε μια οριστική γνώμη σχετικά με τα κριτήρια. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης ε, προτείνεται τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να έχουν ε, τη δυνατότητα όλα αυτά τα θέματα να τα ρυθμίζουν μέσα στην δική τους την ε, επικράτεια ε, με το σύστημα ενός ε, fine tuning ε, το οποίο σύστημα αυτό θα πρέπει να εντάσσεται μέσα σε ένα κοινοτικό πλαίσιο. Και νομίζω, έτσι μπορώ να ολοκληρώσω, ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να πούμε την άποψή μας για αυτή την έκθεση. Δεν πρέπει όμως ούτε να γκρίνουμε ούτε να απορρίψουμε οριστικά τα κριτήρια αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Για να προχωρήσουμε θα πρέπει να γνωρίσουμε επακριβώς τα κριτήρια, όπως επίσης και τις επιπτώσεις τους ε, και την ε, ασφάλεια που προσφέρουν σε σχέση με την επίτευξη του στόχου. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που ήταν ε, ταυτόχρονα σύντομη και ε, περιστατωμένη. Έξι άνθρωποι θέλουν να πάρουν το λόγο. Η κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω για αυτήν την έκθεση και νομίζω ότι τα προτινόμενα κριτήρια ναι μεν αποτελούν μια πολύ καλή βάση για τον ε, διαχωρισμό των μειονεκτουσών περιοχών. Η προϋπόθεση όμως είναι να υπάρχουν τα δεδομένα και να γίνονται προσωμιώσεις, οι οποίες όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Θεωρώ λοιπόν ότι η Κομισιόν καλείται στον ε, τομέα της ε, προσωμείωσης ε, για τα μεμονωμένα κριτήρια να σκεφτεί κάτι διότι δεν είναι, δίκαιο, δεν είναι δίκαια τα κριτήρια αυτά για πάρα πολλές περιοχές σε πάρα πολλούς τομείς ε, όταν είναι ε, κανείς ε, λίγο κάτω από το όριο αυτομάτως απορρίπτεται και αυτό δεν είναι δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για την οριακή τιμή του 66%. Και εδώ τίθεται το ερώτημα γιατί ακριβώς αυτό το ποσοστό Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που θα πρέπει να συζητήσουμε με την Κομισιόν. Όσον αφορά αυτές τις ε, αποχρώσεις, ε, θεωρώ ότι πράγματι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο τομέα, ο οποίος ε, πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί, όπως επίσης και ο τομέας της αυτοδιάθεσης που τον έθιξε ο εισηγητής. Και αυτός προσφέρει την δυνατότητα δικαιοσύνης να επικρατήσει δικαιοσύνη στους διάφορους τομείς. Ευχαριστώ. Κύριος Λάιμ. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή. Νομίζω πως ε, η έκθεση ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο πιστεύω πως και άλλοι ομιλητές ε, σαφώς ε, τόνισαν μέχρι ότου δούμε ποιε είναι οι προσωμιώσει στην εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προσέξουμε πολύ ε, για το αν τελικά να, μέχρι ότου πούμε αν είναι σωστά τα κριτήρια της Κομισιόν. Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με τον αριθμό των κριτηρίων που χρησιμοποίησαν και νομίζω πως υπάρχουν και άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να εξεταστούν και σίγουρα θα προσπαθήσουμε αυτό να το περιμένουμε. Είμαι Εγώ έχω εμπειρία στο θέμα προσωπική. Επίση είναι σημαντικό να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι το μέσο αυτό για να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε ε, ε, γρότες που έχουν υποφέρει από σοβαρό φυσικό μειονέκτημα ακόμα και εκεί που υπάρχουν πολύ σοβαρές ε, προκλήσεις σε σχέση με μειονεκτήματα που έχουν σε σχέση με άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλύτερη υγεία και καλύτερες δυνατότητες για την ε, γεωργία. Πρέπει να επίσης να ενισχύσουμε νομίζω την ε, δυνατότητα εγ, ε, να λάβουμε υπόψη αν τα κριτήρια θα πρέπει να είναι σωρευτικά και να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα ίσως ε, της ε, προσπάθειας αυτής, αλλά το κατόφλι του 66% θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, να δούμε πρώτα τις προσωμιώσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη. Να μας πει και η Κομισιόν πότε περιμένει να πάρει αυτές τις πληροφορίες, γιατί σίγουρα θα μας βοηθήσει για να ενημερώσουμε και αυτήν εδώ την Επιτροπή, να ενημερωθεί μάλλον η Επιτροπή μας, να δούμε κάποιες χάρτες και τη χαρτογράφηση γενικότερα. Σημαντικό θα είναι επίσης εκεί που υπάρχουν περιοχές όπου αφαιρείται γη θα πρέπει να υπάρχουν περίοδοι. Δηλαδή ε, ξαφνικά όταν δει ένας γεωργός να χάνει το 30-40% της γης του δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε μια νυχτά. Θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος μεταβατική για να μπορέσει να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις αλλαγές. Αυτά είναι κάποια στοιχεία και να συγχαρώ τον εισηγητή Ενιγέν για την έκθεσή του. Eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του τον κύριο Ντόρφμαν. Η έκθεση αυτή προϋποθέτει να έχει κανείς ε, κάποιες ειδικέ γνώσεις. Υπάρχει μια κατάταξη σε ενδιάμεσες ζώνες και το κριτήριο της Κομισιόν, ε, η αστιφιλία παραδείγματος χάρη, σωστό είναι αυτό, και επιταχύνει την ε, φυσική υστέρηση. Εξάλλου προωθεί και την ε, αστιφιλία ε, διότι όταν ε, δεν υπάρχει πληθυσμός επιτόπου προάγεται η διάβρωση. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια συμβαστική πρόταση ο πληθυσμός, οι κάτοικοι είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Οι κάτοικοι επιτόπου είναι καθοριστική σημασία και πρέπει κυρίως ε, να λαμβάνετε υπόψη ε, στις ενδιάμεσες ζώνες δεν είναι καθοριστικό κριτήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Κατόπιν, όσον αφορά τη διαχείριση των μειονεκτουσών περιοχών. Αυτό ε, συνήθως συμβαίνει, η διαχείριση γίνεται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Και όταν λοιπόν θα καταρτιστεί αυτός ο χάρτης των ε, μειονεκτουσών περιοχών θα πρέπει να διαβολευτούμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση και θα πρέπει και να ε, διαβουλευτούμε και με τους ε, γεωργικούς συνεταιρισμούς. Ίσως ε, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το ρόλο των γυναικών και να ενισχύσει το ρόλο τους στην τοπική κοινωνία. Ίσως θα πρέπει να ληφθούν περισσότερο οι γυναίκες υπόψη όταν θα καταρτιστεί αυτός ο περίφημος χάρτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ο συνάδελφος, ο κύριος Ντόρφμαν από το νότιο Τυρόλο ε, ανέλαβε την έκθεση. Γιατί ακριβώς επειδή είναι από το νότιο Τυρόλο είναι γνώστης του θέματος και παρουσίασε μια πολύ καλή έκθεση. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα οποία κατέθεσε τώρα η Κομισιόν δεν αρκούν. Δεν είναι δυνατόν όταν ένα από τα οκτώ κριτήρια δεν τηρείται, δεν γίνεται αυτομάτως ολόκληρη περιοχή να χαρακτηρίζεται μειονεκτούσα. Και αν σε ένα κριτήριο ε, το ένα κριτήριο είναι κατά 1% κάτω και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα παραπάνω, αυτά δεν είναι μειονεκτούσα περιοχή. Έχουμε κάνει κάποιους ε, συγκεκριμένους υπολογισμούς και ξέρω, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία αναφέρεται ότι στο Παρίσι, που είναι μία από τις ε, καλύτερες περιοχές της ε, Γαλλίας, εκεί συγκεκριμένες περιοχές ε, καταντάσσονται ως μειονεκτούσες και άλλες περιοχές ορεινές αποχαρακτηρίζονται και δεν είναι πλέον ορεινές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Τι επιδιώκουμε κατ' ουσίαν με την προαγωγή των ορεινών περιοχών επιδιώκουμε να ε, προάγουμε, να προωθήσουμε τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Και δεν είναι δυνατόν με την λάθος εφαρμογή αυτών των κριτηρίων να μην διατηρηθεί η γεωργία στην Ευρώπη, στην έκταση που της αναλογεί. Εμείς ε, ως Κοινοβούλιο που ε, συμμετέχουμε στην συναπόφαση, στη Γεωργία, θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να εκπονηθεί ένας καλός κανονισμός. Έχουμε αρκετό καιρό για να συζητήσουμε και από κοινού ε, με τον κύριο Ντόρφμαν ε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή λύση για να μην υπάρξουν σημαντικά προβλήματα στην Ευρώπη και εμφανιστούν μειονεκτούσες περιοχές που πραγματικά δεν τους αξίζει. Κύριε Σμιτ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Η ενεργός γεωργία σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της, ε, του οικοδομήματος της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εμείς στη Σκοτία έχουμε πολύ καλή εμπειρία με την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ε, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγή θρεπτικών ουσιών και να αντικαταστήσουν άλλα καλλιέργειε όπω παραδείγματος χάρη ο καπνό. Θα είμαι σύντομο. Υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να έχουμε κατά νου. Πράγματι είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να αποφανθούμε οριστικά για την προθέση Κομισιόν γιατί εξακολουθούν να τρέχουν πολλά πράγματα. Και όπω ακούσαμε είναι και το θέμα των αποχρώσεων. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο υπαριθμών 8 για να είμαστε σίγουροι ότι τα κριτήρια αυτά είναι κατάλληλα και ότι οι μειονεκτούσε περιοχέ είναι πράγματι μειονεκτούσε. Μέχρι τώρα είχαμε ε, πρόβλημα με τον κανονισμό. Ήταν περιοχέ ε, στο Λουξεμβούργο που χαρακτηρίζονταν μειονεκτούσε ε, και άλλε που θα έπρεπε δεν τύχαιναν να χαρακτηριστούν. Εμείς θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες για να διασφαλίσουμε ότι η μεταρρύθμιση θα ε, προβληθεί, να ε, είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης και ο προπολογισμός θα πρέπει να υπεραμεινθούμε αυτού ως ένα σωστό τμήμα της πολιτικής ε, για τις λιγότερο ευνοημένες ε, περιοχές. Το να συνδέσει κανείς τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές με την ενεργό κτηνοτροφία, αυτό σημαίνει όμως καταρχήν πρέπει να ορίσουμε τι είναι η ενεργός ε, κτηνοτροφία. στον ορισμό μας των κριτηρίων θα πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε πλήρως και την τοπική αυτοδιοίκηση στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει να πω ότι πραγματικά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή γιατί θέτει το δάκτυλο στους σωστούς ύλου. και αυτά που λέει η Κομισιόν δεν τα κατανοώ Εμεί εδώ και χρόνια προσπαθούμε να προάγουμε τις μειονεκτούσε περιοχές και μιλάμε για το κλίμα και το τι θα κάνουμε με το κλίμα. Εδώ λοιπόν διατρέχουμε κίνδυνο για μένα βλέποντας τα κριτήρια υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και πολύ σωστά τα είπε ο Άλμπερτ. Ε, το γεγονός ότι κάποια κριτήρια ε, καταργούνται από αυτές τις επιδοτήσεις ότι ε, υπάρχει απερίμωση που οδηγεί στη διάβρωση. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό δεν το επιθυμούμε. Συζητήσαμε βέβαια ε, διαμακρών για το θέμα αυτό. Μπορεί κανείς να λέει ότι θέλει για την ενίσχυση του καπνού. Αλλά έχουμε πει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις γιατί είναι μικρές, γιατί προσφέρουν θέσεις εργασίας και γιατί αυτές οι περιοχές πρέπει να παραμείνουν ζωντανές. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα ισχύει γενικότερα για τις ε, μειονεκτούς περιοχές, πόσο μάλλον μάλιστα για αυτές. Και εάν η Κομισιόν έχει ε, πληροφορίες ε, και ξέρει τι έχει επικρίνει το ελεγκτικό συνέδριο, τότε θα πρέπει να δούμε πού ακριβώς εμφανίζεται η κριτική και πώς ακριβώς πρέπει να αλλάξουμε αυτά τα αδύναμα σημεία. Όχι να αναποδογυρίσουμε όλο το σύστημα που εγώ νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούμεθα. Ανατροπής, πλήρους ανατροπής μπορεί βέβαια να κάνω λάθος στην ανάλυση μου. Πάντως εγώ ε, υποστηρίζω ανεπιφύλακτα τον εισηγητή μόνο που εγω νομιζω προς αυτη την κατευθυνση οδηγουμεθα ανατροπης πληρους ανατροπης μπορει να κανω λαθος στην αναλυση μου παντως εγω υποστηριζω ανεπιφυλακτα τον εισηγητη μονο που αυτο το σημείο που σας είπα ε, θα έπρεπε να το προβάλλουμε περισσότερο γιατί όπως παρουσιάζεται τώρα είναι πολύ αδύναμο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να ε, παραμείνουμε στην ε, θέση μας, να προβάλλουμε τη θέση μας. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει επουδενή να μην παραδώσουμε τον δεύτερο πυλώνα στην Περιφερειακή Επιτροπή. Are cuvântul Νίκολσον. Το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φαντάζομαι πως ε, τελειώνει ο χρόνος. Πάντως δεν ήταν το δικό μου το κινητό που φταίει για το μικρόφωνο, σας το πω αυτό. Ε, εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε η Ελίζα Πεθιέγκλε μόλι. Ε, όλοι βασικά λέμε το ίδιο πράγμα. Καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του, για την προσπάθειά του και για το χρόνο του. Ε, εδώ θα πρέπει να προσέξουμε γιατί μπαίνουμε σε πολύ ταραγμένα νερά, επικίνδυνα εδάφη. Ε, μόνο και μόνο επειδή δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο κάνει ερωτήσεις, ε, ε, εμείς θα πούμε, θα απαντήσουμε λέγοντας πόσο ψηλά θέλετε να επιδείξουμε, μα είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται αδρά. 38,5% του μισθού τους έρχεται από εμά. Άρα λοιπόν τον άρχονται και να διαμαρτύρονται για τον κόσμο που ζει στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές ε, και άμα κάθε φορά που ερχόντουσαν μάλλον και μα γκρινιάζαν εμεί συμφωνούσαμε μαζί του και κάναμε το δικό του. δεν θα υπήρχε πια κόσμο στι λιγότερο ευνοημένε περιοχέ. Και συμφωνώ με τον Τζορτ που έφυγε, μέχρι ότου δούμε του χάρτε δεν μπορούμε να έχουμε κάποια άποψη από του θέματο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Επιτροπή να προχωρήσει ούτε καν ένα βήμα ακόμα. Πρέπει να έχουμε τα σωστά κριτήρια και τα σωστά κριτήρια θα πρέπει να ισχύσουν για όλα τα μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο για αυτά που λέει η Κομισιόν. Τα κριτήρια που πιστεύω θα κάνουν μια λιγότερο ευνοημένη περιοχή στην Ισπανία, στην Ελλάδα ή στην Ιταλία θα είναι διαφορετικά από τα κριτήρια που ισχύουν ε, σε περιοχές όπου εγώ ζω, ας πούμε. Και κινδυνεύουμε να κάνουμε ένα κουστούμι one size για όλους εδώ στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να προχωρήσω άλλο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν δούμε του χάρτε. Εμεί θα καταθέσουμε και τροπολογίε και θα συνεργαστούμε με τον εισαγητή. Η Επιτροπή μα, νομίζω, ακολουθεί πολύ λογική προσέγγιση. Αλλά η Κομισιόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μέχρι ότου μα δώσει όλε τι αποδείξει που απαιτούμε, δεν θα συμφωνήσουμε με αυτά που προτείνουν. Ναι. Δεν με νοιάζει. Πού θα τα έρθουν, μπορούν να τα στείλω ήδη στον παρόζο, Α τα πάει και σε πιο ψηλό επίπεδο, αν υπάρχει. Εμεί πάντω θα πολεμήσουμε κατά αυτή τη πρόταση. Ευχαριστώ. Κύριε Μαγκίνη. Σα ευχαριστώ. Άκουσα τι τελευταίε μόνο παρεμβάσει για να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Όπω είπε και ο Τζιμ Νίκολσον, πραγματικά θέλουμε να δούμε αυτέ τι ε, δοκιμέ, να δούμε τι αντίκτυπο θα έχουν αυτά τα κριτήρια στι συγκεκριμένε περιοχέ. Η Ελίζα Πεδιέγκλε το είπε και εκείνη, ότι ορισμένε περιοχέ μπορεί να μην εμπίπτουν για λίγο και ποιε θα είναι οι επιπτώσει για τι εκμεταλλεύσεις σε εκείνες τις περιοχές αν κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και εγώ κλείνω να συμφωνώ για το ελεγκτικό συνέδριο. Ναι, έχουν αναφέρει το θέμα και πρέπει να προσέξουμε για το πώς εμείς αντιδράσουμε στις ανησυχίες που ξέφρασαν. Και επίση να έχουμε στο μυαλό μας τον κόσμο που ζει σε αυτές τις περιοχές. Σήμερα το πρωί παρακολούθησα ε, το θέμα του περιβάλλοντος και την ανάγκη να μείνει κόσμος σε αυτές τις περιοχές και ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να διασφαλίσουμε να έχουν κάποια χρήματα στην τσέπη τους. Και πάλι λοιπόν να συγχαρώ τον εισηγητή και φαντάζομαι πως τώρα δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα του αντίκτυπου και των μελετών αντικτύπου μέχρι το τέλη Φεβρουαρίου. Οπότε έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος είναι ο κύριος Καπούλας Σάντος. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τα όσα ήδη υπόθηκαν να εκτιμήσω, εκφράζω τη θετική μου εκτίμηση για την εργασία του εισηγητή, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να αναφέρω, το 5 και το 8. Εκεί λέει ότι ο εισηγητή στο 5 ότι θεωρεί πω τα 8 κριτήρια που προτείνονται μπορούν να ε, κάνουν, μπορεί να είναι κατάλληλα. Εντάξει, θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα, αλλά θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα και άλλα 8 κριτήρια δικά μα που θα τα σκεφτούμε. Δηλαδή δεν νομίζω πως είναι σωστό να απαριθμώνται τα κριτήρια. Όπως ε, δεν θεωρώ πως είναι θετικό, στο σημείο 8 η πρόταση που κάνει για να χρησιμοποιηθούν οικονομικά στοιχεία. Μα δεν είναι μόνο οικονομικά τα στοιχεία, υπάρχουν και δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ε, συμπεράσματα. Αν βγάλουμε αυτές τις παρατηρήσεις, ε, η έκθεση είναι αξιέπαινη και θα είναι ακόμη καλύτερα αν ο συμπεριλάβει αυτές τις προτάσεις.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 Λοιπόν, να σας πω ότι ορισμένοι τέτοιοι χάρτες υπάρχουν και θα σας ε, πω ε, στη Γαλλία ο χάρτης που επιτρέπει να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα δείχνει πως η Σαμπάνια που είναι μη, που είναι ε, μη ευνοούμενη περιοχή θα είναι ε, μία από αυτές τις μειονεκτικές περιοχές γιατί το 16ο αιώνα τη σαμπάνια τη βρήκανε ε, ως, αντίδοτο στη φτώχεια σε εκείνη την περιοχή. λοιπόν, ε, θα πρέπει δηλαδή να δούμε ποια είναι η φυσική, ποια είναι η πραγματική δουλειά που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε ρεαλιστικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές στον κατάλογο, όπως σας είπα και πριν. Η ε, κυρία Ζωζεφίν Χόμαν αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε να την καλέσουμε να πάρει το λόγο και να είναι σύντομη. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά υπήρξαν πολύ ενδιαφέροντα, πολλά ενδιαφέροντα σχόλια και δεν ε, ξέρω αν θα τα καταφέρω σε ένα λεπτό. Ε, λοιπόν, και εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο, λέει η ομιλήτρια, μάλλον τον εισηγητή εννοεί, γιατί είναι μια εμπεριστατωμένη και ακριβή έκθεση και η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη. Θα ήθελα εξ αρχή να θυμίσω το εξή, που είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Δεν ενεργούμε μόνο επί τη βάση των επικρίσεων του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο ζήτησε και έχει δώσει εντολή στην Κομισιόν το 2005 να αναθεωρήσει τον καθορισμό των λιγότερο ευνοημένων διάμεσων περιοχών, να φτιάξει έκθεση και προτάσεις για το πώς θα γίνει η μεταρρύθμιση του συστήματος. Γι' αυτό το κάνουμε. Διαφορετικά δεν θα είχαμε και τόση δουλειά εδώ. Λοιπόν, αυτή, εδώ, σε αυτό το πλαίσιο δουλεύουμε και επειδή αν μου επιτρέπετε σύντομα θα ήθελα να αποσαφηνίσω τρία σημαντικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν στα σχόλιά σας και θα είναι καλό να τα ξαναδούμε. Καταρχήν, ε, γιατί έχουμε τα κατόφλια. Ε, ο κανονισμός και το σύστημα απαιτούν να υπάρχει ένα σημαντικό φυσικό μειονέκτημα και για να μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο περιοχή υπάρχει σημαντικό μειονέκτημα η το μεγαλύτερο κομμάτι της γεωργικής περιοχής σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να υποφέρει από το ίδιο μειονέκτημα. Αν υπάρχουν όμως έγκυρα ε, ε, γεωργικά συστήματα που πιστεύετε ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν για περιβαλλοντικούς λόγους, μπορείτε να το κάνετε μέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών ε, μέτρων που υπάρχουν. Δηλαδή, τα μέτρα των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, το LFA, δεν είναι το μόνο μέτρο για να παραμείνουν οι γεωργοί και να διατηρηθούν συγκεκριμένα γεωργικά συστήματα σε περιοχές όπου το μεγαλύτερο μέρος της γης δεν εμπίπτει σε αυτό. Ζητήσαμε και για τα κράτη-μέλη και άλλα κατόφλια. Δεν επιμένουμε. Θέλουμε να το ελέγξουν το 66, αλλά μπορούν να, να ελέγξουν και το 50% ή άλλα κατόφλια. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε στο τέλος, όταν θα δούμε τους ε, χάρτες. Και επίσης ζητήσαμε από τα κρατημέλη να μας δώσουν και άλλα κριτήρια, να προτείνουν άλλα κριτήρια, γιατί αναφέρεται συχνά πως πιστεύετε πως αυτά τα κριτήρια δεν μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την Ευρώπη. Και το εξετάσαμε αυτό το θέμα των κρατών μελών και τις προτάσεις τους σοβαρά, μαζί με τους επιστήμονες και το ε, το επιτελείο μας. Τα κριτήρια λοιπόν που αυτή τη στιγμή είναι επιτάπητος μπορούν να θεωρηθούν ως κριτήρια τα οποία είναι αντικειμενικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουμε τι είναι ένα φυσικό μειονέκτημα. Γιατί πιστεύω πως αυτό είναι σημαντικό. Αυτό πρέπει να βγει από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να έχουμε μια σωστή περιγραφή του τι είναι το φυσικό μειονέκτημα για τη γεωργία στην Ευρώπη, υπό διάφορες ε, περιστάσεις βέβαια, με αυτό συμφωνώ αλλά να υπάρχουν κάποιοι γενικοί δείκτες που θα καθιστούν το που θα καθορίζουν μάλλον το πεδίο διακύμανσης των, των φυσικών μειονεκτημάτων στην Ευρώπη. Έπειτα, διατύπωση των κριτήριων, ε, σώρευση μάλλον των κριτήριων. Μπορεί κανείς να σωρεύσει κριτήρια σε, με αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα, μια περιοχή, ας πούμε ιδιαίτερα πετρώδης ή, ιδιαίτερα, ή να έχει πρόβλημα και με το νηφί του εδάφους και με τη θερμοκρασία. Μπορεί να υπάρχει αυτό σε διάφορες περιοχές και ε, φτάνει μέχρι το το 66% του μειονεκτήματος, αλλά έχουμε δυσκολία από την επιστημονική άποψη να δούμε αυτό το μείγμα διαφορετικών κριτηρίων που σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνούν το κατόφλι, δηλαδή το πραγματικό μειονέκτημα όπως αυτό ορίζεται ως εμπόδιο για τη γεωργία. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε να προσθέτουμε ένα μειονέκτημα να φτάνουμε στο 100%, δύο να έχουμε, να με, ή με δύο αν δεν τα καταφέραμε να φτάνουμε στο 60% και ούτω καθεξής. Θα πρέπει αυτό το μέτρο να το δούμε ως μέτρο και μέτρο κατά της ε, απερίμωσης. Ε, είναι ένα μέτρο το οποίο αποφεύγει την εγκατάλειψη της γης. Η διατήρηση του τοπίου είναι μια βασική προϋπόθεση για, ώστε μια περιοχή να μείνει ανοιχτή, κόσμος να κατοικεί εκεί κτλ. Αλλά αλλά για πραγματικά στοχοθετημένη δράση για την παραμονή του κόσμου στις περιοχές αυτές χρειάζονται και άλλα στοιχεία, απασχόληση, συν την ε, προσέγγιση των λιγότερο ευνόμενων περιοχών. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον πληθυσμό για να ορίσουμε τις περιοχές, γιατί και οι πληθυσμοί μετακινούνται με τον καιρό. Εμείς θέλουμε να έχουμε μόνιμα κριτήρια που να μην αλλάζουν. Και τέλος για την ε, καμπανία, το γνωρίζουμε αυτό, ότι αυτό μπορεί να συμβεί, διότι στην καμπανία έχετε πολύ καϊκό έδαφος, πολύ πετρόδες, που όμως ε, τελικά είναι ευνοϊκά, ευνοϊκό για το ειδικό αυτό ποτό που φτιάχνεται εκεί τη σαμπάνια. Αλλά γι' αυτό και έχουμε εισάγει το δεύτερο βήμα τελειοποίησης που υποχρεώνει τα κρατημέλη να φερούν περιοχές με φυσικά με ανεκτήματα τα οποία όμως έχουν ξεπεραστεί λόγω συγκεκριμένης προσαρμογής των γεωργών και των παραγωγών τους που ξεπερνούν το μειονέκτημα. Η καμπανία λοιπόν δεν θα είναι στο χάρτη αν το κράτος μέλος έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, κύριο Ντόφμαν, για τις τελευταίες του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, αυτά που ελέγχθησαν ακολουθούν όλα την ίδια κατεύθυνση και κατόπιν τούτου δεν έχω κι εγώ πολλά να προσθέσω. Ε, τέθη το θέμα του facing out. Ε, σωστό αυτό. θα υπάρξει μετατόπιση περιοχών και πρέπει να εξετάσουμε κυρίως το θέμα εκείνων των περιοχών που θα αφαιρεθούν από όλο αυτό το σύνολο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχω την, ε, κατά νου την τελευταία παρατήρηση όπου επισημάνθηκε ότι πολλές φορές η στέρηση έχει σχέση και με την καλλιέργεια. Στη συγκεκριμένη περιοχή, στην Καμπανία, εκεί έχουμε μία καλλιέργεια η οποία διατηρείται ε, ακριβώς ε, γιατί υπάρχει αυτή η αυτό το μειονέκτημα. Ε, το στον Μπορντό, ε, παραδείγματος χάνει, ισχύει το ίδιο. Αν στον Μπορντό, παραδείγματος χάνει, καλλιεργήσει κανείς σιτηρά, θα πρόκειται για καταστροφή. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απόλυτο αυτό που αναφέρετε για τις ε, καλλιέργειες. κάπως θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση για αυτό το περίφημο fine tuning. Και επιτρέψτε μου και δύο λόγια για τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ο κανονισμός ε, στον στον οποίο βασίζονται όλα αυτά, ε, αποκλείει τα οικονομικά κριτήρια. Εγώ στην έκθεσή μου ε, προσπαθώ να ξαναθέσω το θέμα μέσα από το fine tuning γιατί θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι λογικό. Ε, το να ε, συμπεριληφθεί η τοπική ε, περιοχή αυτό έχει οδηγήσει στο ότι είχαμε τελικά μέχρι τώρα πολύ καλές εκθέσεις και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε αυτή η συμπερίληψη. Κατόπιν υπάρχει και ένα άλλο κέριο θέμα που ετέθη. Πώς ακριβώς μπορούμε να βρούμε τις σωστές περιοχές. και αυτό είναι ένα κέριο θέμα όπως σας είπα ε, είναι και ένα θέμα σημαντικό, πολιτικό ε, οι ε, καλλιεργητές πρέπει να γνωρίζουν το σύστημα και να νιώθουν ότι το σύστημα είναι δίκαιο κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα θα ήθελα ε, θερμά να ευχαριστήσω ε, κυρίως ε, τους συνεργάτες στην Κομισιόν αλλά και στη Γραμματεία και βεβαίως χαίρομαι πάρα πολύ που τις επόμενες εβδομάδες θα δεχθώ τις βελτιωτικές προτάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία ε, είναι 4 Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα και η ψηφοφορία ε, θα γίνει στις 16 και 17 Μαρτίου ε, και στην Ολομέλεια του Απριλίου. Συνεχίζουμε. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση ε, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγητής, ε, συντάκτης γνωμοδότης είναι ο κύριος Καρόνα και ε, του δίνω το λόγο. Mm, το μικρόφωνο έχει κάποιο πρόβλημα, θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει η έκθεσή μου που έχει μεταφραστεί σε όλες τις ε, γλώσσες και βλέποντας την προκεχωρημένη ώρα, εγώ δεν θα χρειαστώ πάρα πολύ για να σας πω ε, ταχύτατα θα έλεγα να θίξω ορισμένα θέματα επί της ουσίας που αφορούν σε αυτό το έγγραφο. Το πρώτο λοιπόν θέμα, κατά την άποψή μου, ουσιώδους ε, σημασία που προσπάθησα να το συμπεριλάβω στη γνωμοδότησή μου αφορά στο ότι είναι απολύτως απαραίτητο να διαχειριστούμε τα βιολογικά απόβλητα και αυτό μέσα από έναν φυσιολογικό κύκλο που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων τόσο όσον αφορά την διαφύλαξη των ε, πρώτων υλών όσο και την μείωση της, των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Υπάρχουν λοιπόν δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, και είναι σαφή πάνω από το 41% των οργανικών αυτών αποβλήτων εναποτίθενται σε χωματερές. Κατόπιν τούτου, όσον αφορά την, ε, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά σε όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι εύκολα μπορείτε να τα κατανοήσετε. Κατόπιν τούτου, η, ε, η διαχείριση σε χωματερές σε ανοιχτούς χώρους διάθεσης είναι μια λύση αλλά δεν είναι η καλύτερη και ε, λαμβάνεται υπόψη μόνο ως έσχατη λύση. Κατόπιν τούτου η δική μας η προσπάθεια και την εκφράζουμε αυτή και στη γνωμοδότησή μας είναι να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις με τις οποίες θα μπορέσουμε την επιλογή μας να την ε, καταστήσουμε την ε, καλύτερη και η λύση των χωματερών να μην χρησιμοποιείται η δυνατόν. Το θέμα λοιπόν το οποίο εξετάζουμε και στη γνωμοδότησή μας, το θέμα της πρόληψης. Αυτό βεβαίως είναι το πρώτο καθοριστικό στοιχείο στον αγώνα που διεξάγουμε και στην ιεράρχηση των αποβλήτων. Εγώ Όσον αφορά την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, ε, γνωρίζουμε ότι το μέλλον της ε, γεωργίας εξαρτάται και από τις ε, πολιτικές διαφύλαξης του εδάφους. Έτσι λοιπόν η κομποστοποίηση και η αναρεόβια διαχείριση θα μπορούσαν να αποτελούν μια εναλλακτική λύση στη χωματερή και διότι μέσα από αυτό το σύστημα μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση της γονιμότητας των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Η μέθοδος λοιπόν της ε, συγκέντρωσης ε, των αποβλήτων αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα η ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κομπόστ αυτή η ποιότητα χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα του τελικού προϊόντος πολύ έτσι ενδεικτικά θα ήθελα να σας πω ότι για αυτούς ακριβώς τους λόγους καλέσαμε την Κομισιόν να αναζητήσει δεσμευτικούς την ε, οριοθέτηση δεσμευτικών στόχων όσον αφορά την ανακύκλωση και που θα ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και κλείνω με αυτό να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή τα απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μιλάμε για 66 μέχρι 102 εκατομμύρια τόνους. Μιλάμε για έναν τέτοιο όγκο αποβλήτων που προκύπτουν από την βιομηχανία των τροφίμων και των ποτών. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και ε, επειδή βεβαίως δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και νομίζω ότι ε, τελικά όλοι μπορέσατε να δείτε τη δική μου τη γνωμοδότηση ε, περιμένω τις τροπολογίες σας για να μπορέσω και εγώ να καταλήξω σε μια όσο πιο καλή έκθεση που θα συμβιβάζει τις διάφορες απόψεις. Σας ευχαριστώ κύριε Καρόνα. Όντως, εξαντλήσαμε το χρόνο μας. Οι παρεμβάσεις θα είναι μονόλεπτες, γιατί διαφορετικά θα κρατήσουμε του ήρμηνε. Ναι, υπόσχομαι, είμαστε όλοι κουρασμένοι, θα μιλήσω πολύ λίγο. Να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, δουλειά του, για αυτή την έκθεση. Εγώ έχω κάποιε προτάσεις που ελπίζω θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια συμβαστική. Έχω δύο σχόλια. Το ένα αφορά μια ανησυχία που έχω ότι η κομποστοποίηση θεωρείται ω λύση για τα προβλήματα, για τα εδάφη, γιατί ο όγκος ε, λιπάσματος που μπορούμε να φτιάξουμε και η γη που μπορεί να καλύψει είναι πολύ μικρή. Έχει σχέση αλλά ίσως να μην είναι τόσο έντονη Επίσης οι γεωργικές ε, γες, οι αρρώσιμες γες να μην ε, καταλήξουν να είναι χωματερές ας πούμε για κακής ποιότητας λιπάσματα. Και έπειτα, ε, ίσως να μην είναι δικό μας θέμα να το συζητήσουμε, αλλά να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το σύστημα ε, των υπονόμων για να παίρνουμε και απόβλητα τροφίμων. Τώρα, αυτοί που ζουν ε, κοντά στις χωματερές είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να συνηθίσει και την ιδέα. Αν δεν δεχτούμε την κομποστοποίηση θα πρέπει να δεχτούν την ιδέα ότι θα υπάρχουν τέτοιου είδους δυνατότητες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια συγκεκριμένα μέρη ε, όπου θα γίνεται η κομποστοποίηση. Θα, θα, είναι περισσότερα από ό,τι χωματερές. Εν πάση περιπτώσει θα υποβάλω κάποιες σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε κύριε Σιγητά για τη γνωμοδότησή σας και θα ήθελα απλά να κατευθύνω σαφές ότι σε αυτόν τον τομέα ε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν νομοθετικές διατάξεις και θα υπάρξουν μόνο αν πραγματικά οδηγήσουν σε αποτελεσματική διαχείριση και όχι απλά και μόνο για να υπάρξουν νέα γραφειοκρατικά προσκόμματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να συζητήσουμε για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας γιατί ε, στη Γεωργία η διαχείριση των αποβλήτων έχει μεγάλη, ασκεί μεγάλη επιρροή στην ποιότητα του εδάφους, ε, στα ύδατα, στην γονιμότητα και στην ε, δέσμευση του άνθρακα. Εγώ προσωπικά το βρίσκω σωστό που επισημαίνει ο κύριος Εγκαρόνα ότι η αναπόθεση σε χωματερές είναι η τελευταία η έσχατη λύση ε, γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Κατόπιν τούτου τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει να καίγονται μόνο εφόσον μπορούν να ε, αποφέρουν κάτι για την εξοικονόμηση και ε, απόκτηση ενέργειας. Αλλά και αυτό πάλι είναι έσχατη ε, λύση. Στη Γερμανία υπάρχει ήδη ένας κανονισμός σχετικός. Εμείς έχουμε πολλά βιολογικά απόβλητα και νομίζω ότι στον τομέα αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε υποδειγματική στάση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι δεν ε, μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια να, εξακολουθήσουμε να αποθέτουμε τα απόβλητα στις ε, ανοιχτές χωματερές που ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Και η καύση είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. Ε, μπορεί να αφορά μόνο κάποια ε, στοιχεία των βιοποβλήτων. Εμείς πιστεύουμε καλύτερα να γίνεται εκμετάλλευση μέσα από το βιοαέριο, κυρίως ε, σε απόβλητα από τα τρόφιμα ε, σήμερα αυτό από πλευράς τεχνικής δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, είχαμε μεγάλο άλμα στην τεχνολογία Και θα μπορούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε ενδεχόμενο όλα αυτά να τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν με βιοαέριο. Η Κομισιόν λοιπόν εκπροσωπείται με την κυρία Φράς. Παρακαλώ. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Σας παρακαλώ ένα λεπτό το πολύ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες για όλα αυτά τα πολύ ε, έγκυρα σχόλια τα οποία σημείωσα για να τα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Εμείς θέλουμε να καλωσορίσουμε το ενδιαφέρον στο ντοσχέ αυτό και την εξέταση του από την Επιτροπή. Εκτιμούμε τη λεπτομερή ανάλυση του ντοσχέ και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Υπήρξαν διάφορα θέματα τα οποία είχαν αναφερθεί στο πράσινο βιβλίο. Βλέπω πως έχουμε κοινέ απόψεις και παρόμοιες ε, ε, θέματα προσυζήτηση σε περίπτωση που αποφασίσουμε να ενεργήσουμε στον τομέα αυτό. Ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω κάποια σημεία τα οποία ε, με χαρά σημειώνουμε σε αυτή την, το σχέδιο γνωμοδότησης, δηλαδή η στήριξη στο θέμα της ιεραρχίας των αποβλήτων και η πρόληψη, η υποστήριξη για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, καθώς και η απαγνώριση των βιοεποβλήτων ως, ένα, ως πολύτιμη πηγή ε, και πόρο, ε, την χρήση των ε, λοιπασμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας των γεών και την ανάγκη για ποιοτικές, ποιοτικές προδιαγραφές. Προσβλέπουμε λοιπόν στην τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής σας για την ε, ε, έκθεση μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε κύριε Καρόνα να, να μας αναφέρετε τα συμπεράσματά σας, τα τελικά. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και δεν μπορώ να πω στην ουσία, αλλά θεωρώ ότι από αυτά που κατάλαβα, όλα αυτά που ελέγχθησαν εμπλουτίζουν, εξειδικεύουν, ε, καθιστούν ακόμα πιο ε, πιστική την έκθεση που σας ε, παρουσίασα. Εγώ λοιπόν τις ευθύς τις αμέσως επόμενες ημέρες περιμένω τις τροπολογίες έτσι ώστε να μπορέσω όπως σας είπα να δώσω σε αυτήν την έκθεση μια όσο πιο ομοιόμορφη θέση γίνεται που να εκπροσωπεί την ε, Επιτροπή μας. Πρόεδρος, η καταλεκτική ημερομηνία ε, για τις τροπολογίες 2 Φεβρουαρίου και θα ψηφίσουμε στις 22 Φεβρουαρίου το 2010. Στα διάφορα έχω μόνο μία ανακοίνωση να σας κάνω. Εχθές το απόγευμα οι συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων αποφάσισαν να επιβεβαιώσουν την έκθεση Κέρσκι που αφορά στις ε, ενισχύσεις για λιγότερο ευνοημένες περιοχές ε, και θα προτείνουμε στην Ολομέλεια αυτό να ψηφιστεί το Μάρτιο του 2009 ε, κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης. Και αν δεν έχετε αντιρρήσεις θεωρώ ότι εγκρίνεται η πρόταση αυτή και η επόμενη συναντησή μας θα λάβει χώρα